Πρόκειται για μια συνωμοσία. Κατ' ουσίαν ναι, τίποτα δεν είναι καινούριο. Αυτή είναι μια παλιά ιστορία η οποία απλά ε, εφαρμόζεται στη νέα τεχνολογία της ε, τεχνητής νοημοσύνης. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν ε, από όλα αυτά να βγάλουμε νόημα γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε και να κατανοήσουμε πού ακριβώς κατευθυνόμαστε. Υπάρχουν δύο ιστορίες πάρα πολύ καλές και είμαι πολύ ευτυχής και για τις δύο. Η μία είναι γιατί τελικά τα καταφέραμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ ε, δουλεύω πάνω σε αυτό το μοντέλο εδώ και 20 χρόνια και άλλοι δουλεύουν πολύ περισσότερο. Ε, επιτέλους συμβαίνουν αρκετά πράγματα μετά από μια τεράστια επένδυση και την ίδια στιγμή έχουμε ε, μία παγκόσμια υποδομή δεδομένων που τη χρησιμοποιούμε. Αυτά τα δύο πράγματα κατ' ουσίαν ε, αλληλοσυνδέονται και το ένα άλλο συμπληρώνει το άλλο με καταπληκτικό τρόπο. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι συμβαίνουν ε, πάρα πολλά γεγονότα που εξηγούν κατά κάποιον τρόπο το τι ακριβώς βιώνουμε. Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά τους. Τι ακριβώς είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, μέχρι τη δεκαετία του 90, οι άνθρωποι πίστευαν ότι η σε συμπεριφορά ε, προέκυπτε από την ε, λογική και από μηχανές ε, οι οποίες σκέπτονται με βάση κανόνες που είναι γνωστοί καταρχήν στο σχεδιαστή. Έτσι λοιπόν για μένα που είμαι ο ειδικό της ε, ε, τεχνητής νοημοσύνης. Ε, το σκάκι είναι πολύ σημαντικό. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα και έτσι κάποια στιγμή κατασκευάσαμε μηχανές που θα μπορούσαν να σκεφτούν. Πάντως, για δεκαετίες ολόκληρες επενδύσαμε στο να κατασκευάσουμε μηχανές που σκέφτονται λογικά, που γνωρίζουν γεγονότα και πιστεύαμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να έχουμε όραμα, μετάφραση, ρομποτική πλοήγηση, αναγνώριση ήχου. Σήμερα όμως ε, μιλάμε για αυτοκίνητα που πηγαίνουν μόνα τους, ε, ε, για το translate της Google και όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν, είναι το αποτέλεσμα μιας συνέλευσης που είχε ξεκινήσει το 1958. Όλα αυτά τότε ε, τα σκεφτήκαμε και κατέστησαν δυνατά πρόσφατα. Έχουμε λοιπόν συστήματα που σκέπτονται λογικά για γεγονότα και όλα αυτά έγιναν με πολύ διαφορετικό τρόπο που είναι πολύ σημαντικός για μας. Ο τρόπος με τον οποίο ασχολούμεθα σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι συγκεντρώνοντας παραδείγματα της συμπεριφοράς που θέλουμε να αναπαράγουμε. Θέλουμε δηλαδή ε, πολλά παραδείγματα της μεταγραμμένης ε, γλώσσας ε, και μάλιστα η δική μου ομιλία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει Επίσης ε, είναι ότι έχουμε έναν αλγόριθμο ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει τη συμπεριφορά μιας ε, μηχανής. Αυτό λοιπόν το κομμάτι του ε, αλγορίθμου μάθησης, ακριβώς αυτό το κάνουμε εδώ και 20 χρόνια. Και αυτό ακριβώς δημιούργησε τα πάντα. Σήμερα λοιπόν έχουμε την AlphaGo, την PlayGo, ε, τα Google Cars, όλα αυτά ε, έχουν, ε, τα έχουμε μάθει από την εμπειρία, τα φίλτρα, τα φίλτρα σε spam. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορούμε να παραγγείλουμε βιβλία, να έχουμε μεταφράσεις από αλγορίθμους όλα αυτά ε, που μπορεί να μην μοιάζουν με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είναι κάτι το οποίο κατέστη ε, δυνατό τις ε, τελευταίες δεκαετίες. Και παλαιότερα αυτά ήταν απλά ένας εκπαιδευτικός στόχος. Πώς φτάσαμε λοιπόν, φτάσαμε εδώ μέσα από την εκπαίδευση. Ε, σήμερα αυτό που ε, έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι η ε, κόμισα του ε, η οποία παρατίθεται, ήταν λάθος. Αυτή παρατίθεται και, λέει, έλεγε ότι οι μηχανές κάνουν πράγματα που μπορεί κανείς να τα εξηγήσει, αλλά η δική μου, οι συνάδελφοι που κατασκεύασαν την AlphaGo στο Λονδίνο, δεν μπορούν να το να εξηγήσουν, αλλά το κατασκεύασαν. Οι μηχανέ μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν και που πρέπει να τα εξηγήσουμε. Αυτό έχει σχέση με τη μηχανική μάθηση και αυτό ε, θα είναι και σημαντικό αργότερα. Δηλαδή, οι μηχανέ κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν. Οι ε, intelligent agents πολλές φορές προκύπτουν από συσχετισμούς, συσχετισμοί που εντοπίζονται στα δεδομένα. Και αυτό βέβαια δεν εξηγεί το φαινόμενο. Αν θέλω να σας συστήσω ένα βιβλίο, μπορώ να κάνω συσχετισμούς με την ιστορία σας. Ε, δεν ξέρω βέβαια αν θέλετε να αγοράσετε αυτό το βιβλίο. Ε, θα πρέπει να μάθω την προσωπικότητά σας, ε, τα γούστα σας. Το ίδιο ισχύει και για την AlphaGo και για πολλά άλλα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι μια επιστημονική ανακάλυψη που έλαβε χώρα τα τελευταία χρόνια και αυτό δεν το αναγνωρίζουμε ως ε, επιστήμη. Η συμπεριφορά των ανθρώπων μπορεί να προβλεφτεί απλά και μόνο με συσχετισμούς ε, σε σχέση με την ε, παρελθούσα συμπεριφορά τους. Δηλαδή μπορούμε να προβλέψουμε το τι θα γίνει σε παρεμφερείς καταστάσεις και αυτό για πολλούς ανθρώπους απλά ρίχνοντας μια ματιά στην παρελθούσα συμπεριφορά τους. Βεβαίως αυτό ε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να νικήσει τις ε, μηχανές που ε, ασχολούνται με τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Έχουμε ένα βιβλίο πολύ δημοφιλές για τα big data και ακριβώς εκεί αναφέρεται ότι οι συσχετισμοί υπερισχύουν των προκλήων και των αιτίων κυρίως όσον αφορά στα δεδομένα. Και τα δεδομένα υπάρχουν παντού. Και αυτό είναι το άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Ε, αυτό τώρα που ζούμε είναι σαν είναι μια νέα μορφή πετρελαίου. Θα σας αναφέρω πολύ σύντομα ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα βαθμολόγιο όπου εντάσσονται διάφοροι πόντι, διάφοροι βαθμοί και με βάση αυτό μπορεί κανείς να ανατρέξει στο παρελθόν. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως όσον αφορά φάρμακα που δίδονται σε ασθενείς. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς γιατί, αλλά το, η συγκεκριμένη εταιρεία με βάση τα δεδομένα που συγκέντρωσε μπόρεσε να κάνει ακριβώς αυτό τον ε, συσχετισμό ανάμεσα στις διάφορες μεταβλητές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ασθενών και μπόρεσε να φτιάξει και έναν κατάλογο με προβλέψεις Αυτό λοιπόν δείχνει ότι είναι ένα παράδειγμα μιας ε, μητέρας, με ανήπαντρης μητέρας, η οποία θα ε, χρησιμοποιούσε, τα έπαιρνε περισσότερα και πιο συχνά φάρμακα αν τις δινόντουσαν κουπόνια. Αυτές είναι κάποιες πληροφορίες που μπορούμε να συγκεντρώσουμε, δεν τις κατανοούμε, απλά γίνεται ένα συσχετισμός. Και τα δεδομένα παρεπιπτόντως μπορεί κανείς και να τα αγοράσει. Και τα ίδια δεδομένα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να κάνει εκλογικές προβλέψεις και παρεμφερία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς μπορεί κανείς να μιμηθεί την ανθρώπινη συμπεριφορά και να την παρουσιάσει, να την αναλύσει αν έχει τα απαραίτητα δεδομένα. Πριν από κάποια χρόνια όλοι μιλάγανε για τα δεδομένα, όπως σας είπα, για τη νέα μορφή πετρελαίου. Δηλαδή μια οικονομία που θα βασίζεται στα δεδομένα στην Ευρώπη. Τα δεδομένα, τα data, ήταν αν θέλετε η λύση για τα πάντα. Και με τον τρόπο αυτό προέκυψαν πολλές προσδοκίες. Και έτσι φτάνω στο δεύτερο σκέλος της ομιλίας μου. Πώς θα συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Γιατί αν θέλουμε να έχουμε ένα τέτοιο ευφυές σύστημα, θα μπορούσαμε να το παράγουμε, αλλά πού θα βρούμε όλα αυτά τα δεδομένα. Και αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα. Πώς μπορεί κανείς να συγκεντρώσει όλα αυτά τα δεδομένα, έτσι ώστε να προβλέπει τη συμπεριφορά των ανθρώπων ε, να γνωρίζει αν θέλετε τις συνθιές τους, ε, στο, τι διαβάζουν. Αυτό τώρα είναι κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Κατά το παρελθόν ε, είχαμε τη συγκεκριμένη υποδομή των ε, τηλεφώνων, ε, των τραπεζών, των, της αλληλογραφίας Τώρα όμως ε, η υποδομή είναι τελείως ε, διαφορετική και τα τελευταία 20 χρόνια έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος η οποία αντικαθιστά την παλαιότερη υποδομή. Έχουμε ένα νέο μέσο και αυτό το νέο μέσο τώρα πλέον μπορεί να κάνει αγορές, ε, να προσφέρει ψυχαγωγία, πληροφορίες. Πώς μπορούμε λοιπόν να φτάσουμε στο ίδιο σημείο με την ίδια υποδομή. Αυτό είναι σημαντικό. Ένας βασικός παράγων που κατ' ουσίαν μελετήθηκε σε βάθος ήταν ότι μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τους ενδιάμεσους, να τους παραγωνίσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πριν από τον ιστό υπήρχε κατ' ουσίαν ε, δίναμε ιδιαίτερη σημασία στους φρουρούς. Αυτοί ε, που είχαν τα κλειδιά, ας πούμε, των μέσων ενημέρωσης, δηλαδή ένας πολιτικός για να εκλεγεί θα έπρεπε να έχει πολύ καλές σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης. Ή οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές ε, στις μουσικές βιομηχανίες. Αλλά και εσείς, αν θέλετε να κλείσετε κάποιο ταξίδι, θα έπρεπε να απευθυνθείτε σε γραφείο ταξιδίων. Πώς θα μπορούσατε να διαφημιστείτε, να πάτε σε μια διαφημιστική εταιρεία. Όλοι αυτοί ήταν φρουροί, όπως τους αποκαλούμε οι ενδιάμεσοι, εκείνοι οι οποίοι βρισκόντουσαν στη μέση της ε, αλυσίδας αξιών της οικονομίας. Και αν θέλει κανείς να γνωρίζει πώς μοιάζει ένας τέτοιος ε, φρουρός που έχει τα κλειδιά. Ε, υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κρατάνε τα κλειδιά και ελέγχουν τα πάντα και κάποια στιγμή ε, αρκετοί πίστεψαν ότι πρέπει να υπάρχει μια υποδομή που θα επιτρέπει να πολλούνται τα προϊόντα κατευθείαν από τον παραγωγό στον καταναλωτή, από τον εκδότη στον αναγνώστη. Αυτό λοιπόν ήταν η στιγμή της απελευθέρωσης. Πελευθερωθήκαμε από τους ενδιάμεσους και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την οικονομία, τη δημοκρατία, την κοινωνία. Αυτή η κατάργηση των ενδιάμεσων ήταν ένα βήμα προς ε, μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό, να μην υπάρχει έλεγχος από τους ενδιάμεσους, αλλά η εξουσία απευθεία στο λαό. Αυτά όταν ε, πρωτοπροέκυψε ο ιστός στο διαδίκτυο. Αυτή ήταν μια μεγάλη υπόσχεση και νομίζω ότι στην αρχή, στην αρχή αυτής της επανάστασης επιτέλους ε, είδαμε ε, ότι υπάρχουν αυτά τα βίντεο, αλλά πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχαν. Είχαμε τους καταγγέλλοντες, θα τα μαθαίναμε όλα αυτά, ακόμα και συγκρίνοντας ε, τιμές, να ξέρουμε ας πούμε ποια είναι, ποιο είναι το πιο φθηνό δωμάτιο που υπάρχει ε, σε αυτή την πόλη ή ο ανταγωνισμός μεταξύ των ανθρώπων. Αυτά μπόρεσαν να λειτουργήσουν, ήταν πίσω από τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και εμείς τα υιοθετήσαμε, εξοικονομήσαμε χρήματα, αποκτήσαμε μεγαλύτερη αυτονομία και μπορέσαμε να αντικαταστήσουμε πολλές δομέ εξουσία. Και αυτή είναι μια μεγάλη επανάσταση που έφερε το διαδίκτυο. Δέστε λοιπόν εδώ, μπορείτε να συγκρίνετε τιμές στο κινητό σας για προϊόντα, για ξενοδοχεία, για τις ε, ειδήσει. Μπορείτε και να τους αναγκάσετε να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, να ε, επιφέρετε ακριβώς το αντίθετο, να αντιστρέψετε την εξέλιξη, να τα κάνουν όλα αυτά για εσάς. Και όλες αυτές τις πληροφορίες τις έχετε στο κινητό σας. Στην αρχή αυτή ήταν η μεγάλη μας ελπίδα. Αυτό θέλαμε παράλληλα ε, καθώς ε, κάνετε την ε, επιλογή σας τους δίνετε κάποια δεδομένα δηλαδή ποιο ξενοδοχείο επιλέγετε πότε, ποια στιγμή της ημέρας το κάνατε αυτό, πόσα χρήματα πληρώσατε άρα η εταιρεία που προσφέρει την υπηρεσία παίρνει κάποια προμήθεια από τη συνολογή αλλά και παίρνει και κάποια δεδομένα που μπορεί να τα αναλύσει αν θέλετε είναι μια συναλλαγή δίκαιη Μερικές φορές μάλιστα αυτές οι εταιρείε δεν παίρνουν καν προμήθεια, θέλουν μόνο τα δεδομένα. Άρα δηλαδή ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο, το να παίρνει κανείς προμήθειες ή το να παρατηρεί τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Αυτά τα δεδομένα όμως είναι εκείνα που κατέστησαν δυνατή την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι μπορέσαμε να καταλήξουμε στο πώς μπορεί κανείς να καταργεί κάποια μέλη στο spam. Ε, προέκυψε λοιπόν μια νέα υποδομή που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή την υποδομή δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε στα χέρια μας χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δηλαδή το πρώτο βήμα. Δεν μπορεί κανείς ε, να χρησιμοποιεί μια βιβλιοθήκη με ένα εκατομμύριο βιβλία αν δεν έχει ε, την κατηγοριοποίηση. Δεν μπορεί να διαβάσει ε, κανένα βιβλίο ή να δει ένα βίντεο αν δεν έχει μία μηχανή αναζήτησης που βοηθάει να βρει κανείς αυτό το βίντεο. Δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονος κόσμος χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη και δεν μπορεί να υπάρξει τεχνητή νοημοσύνη αν δεν υπάρχει το δίκτυο το οποίο αναλύει και ε, αναλύει τη συμπεριφορά των ανθρώπων και καταθέτει προτάσεις. Άρα δηλαδή το σύστημα άρχισε να αυτοτροφοδοτείται και έτσι ε, πολύ γρήγορα επιταχύνθηκε όλη αυτή η διαδικασία. Όλα αυτά λοιπόν τα μαζικά δεδομένα πολύ γρήγορα έγιναν προσπελάσιμα και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε πρόοδο στην τεχνητή νομοσύνη. Γιατί έχουμε τα δεδομένα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτές λοιπόν οι δύο εφευρέσεις ε, συνδυάστηκαν και πρόκειψε ένα όνομα για τα δεδομένα που μπορούσαμε να λύσουμε Μιλάμε data in the wild, έτσι τα αποκαλούμε. Δηλαδή υπήρχαν αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να τα αναζητήσουμε, ε, Παραδείγματο χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη ε, μπορεί να γίνει κάποια ευφυής μετάφραση ε, γιατί υπάρχουν τα δεδομένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν data in the wild όπως τα λέμε αλλά μπορεί κανεί να τα χρησιμοποιήσει και σε συζητήσεις υπάρχουν θέλετε και τα like και αυτά δίνουν δεδομένα ή το να βλέπει κανείς κάτι στα, στην τηλεόραση, στο κινητό όλα αυτά είναι δεδομένα τα τελευταία χρόνια όλοι μιλάνε για δεδομένα, την επιστήμη των δεδομένων, big data, το, ε, τη νέα, το νέο πετρέλαιο, data in the wild. Βλέπουμε ότι προκύπτει νέο υλικό επιτρέποντας τις εταιρείες να ε, συγκεντρώνουν τα στοιχεία μας. Αυτή ήταν μια άρρητη συμφωνία που προέκυψε. Δώστε μας λοιπόν αυτό που έχετε να προσφέρετε και εμείς ε, θα σας δώσουμε τα δεδομένα μας. Αυτή ήταν η συναλλαγή και όλα πήγαιναν καλά, το σύστημα λειτουργούσε, εξακολουθεί να λειτουργεί, ε, μας βοηθάει στο να έχουμε μεγαλύτερη αυτονομία. Μέχρι που μία ημέρα όταν αρχίσαμε να βλέπουμε κάτι τέτοιο και εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα οι άνθρωποι ξεπλάγησαν για δέστε το λιγάκι. Βλέπουμε ότι υπάρχει ε, μία τράπεζα δεδομένων στην NSA, ε, στην Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ. Η Wikileaks ισχυρίζεται ότι ε, η CIA μπορούσε να παρακολουθεί με τα κινητά και να τοποθετεί κοριούς, πάρα πολλές τέτοιες πληροφορίες. Οι άνθρωποι λοιπόν άρχισαν σιγά σιγά να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται ναι, μεν ε, καλωσορίζουμε ή χαιρετήσαμε αυτή την τεχνολογία στην καθημερινή μας ζωή, τώρα όμως για πρώτη φορά προέκυψαν πράγματα που δεν μας άρεσαν και σκεφτήκαμε για πρώτη φορά δεν τα θέλουμε αυτά. Παρεπιπτόντως, εγώ δεν νομίζω ότι όλα αυτά ήταν και απρόσμενα, έτσι και για να είμαι και ειλικρινής. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα, στο Guardian ε, στην ισοσελίδα της Guardian ε, δημοσιεύτηκε αυτό που βλέπετε και εδώ αναφέρεται ότι όλες αυτές οι εταιρείε μπορούν να προσφέρουν δεδομένα στις υπηρεσίες ασφαλείας. Δεν ε, το επιβεβαιώνω, απλά το ισχυρίζεται αυτό ο Guardian. Και οι άνθρωποι σοκαρίστηκαν όταν το άκουσαν αυτό. Μα πώς ήταν δυνατόν να περιμένουμε κάτι άλλο τη στιγμή που όλα μας τα δεδομένα τα δίνουμε σε ένα μοντέλο και τα στέλνουμε σε μια γραμμή επικοινωνίας που δεν ελέγχουμε. Όποιος κατανοεί λιγάκι την ιστορία θα γνωρίζει πολύ καλά ότι ε, θα μπορούσε κάποιο να αγοράσει ένα μεγάλο δίσκο και να τα αποθηκεύσει αυτά τα δεδομένα. Ούτε και εμένα μου άρεσε η εξέλιξη, αλλά δεν εξεπλάγει. Πάντω, όταν προέκυψαν όλα αυτά, οι άνθρωποι άρχισαν να σκέπτονται και σκέφτηκαν κάτι πολύ σημαντικό. Ότι πλέον δεν μπορούσαν, δεν είχαν οδό δρόμο διαφυγή. Ε, εγώ σκέφτηκα ότι ε, δεν θα αγοράζω πια το ε, κινητό μου, θα έχω τηλεφωνικό κατάλογο, δεν θα το παίξω αυτό το παιχνίδι. Κάποια μέρα όμως διαπιστώσαμε ότι δεν γίνεται αυτό. Αυτά λοιπόν ε, συνέβησαν και κατά κάποιον τρόπο ξυπνήσαμε. Δεν μπορούμε πλέον να λειτουργήσουμε αν δεν είμαστε ένα μέρος του συστήματος. Όμως το σύστημα ελέγχει τις δραστηριότητε μας και αυτό δεν μας αρέσει. το Βεβαίω, ε, δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη λύση, αλλά η μαζική εποπτεία, ο μαζικός έλεγχος, ε, κατ' ουσίαν δεν είναι και το τέλος ιστορίας, δεν τελειώνει εκεί η ιστορία. Συνέβησαν και πάρα πολλά άλλα καινούργια που εξηγούν γιατί οι άνθρωποι τώρα ανησυχούν ακόμα πιο πολύ. Τελικά, αν κάτι είναι νόμιμο και αποφέρει και κέρδη, κάποιος θα ασχοληθεί. Έτσι λοιπόν, αν η συγκέντρωση και εκμετάλλευση δεδομένων μπορεί να γίνει νομικά και να αποφέρει και χρήματα, προφανώς οι άνθρωποι θα ασχοληθούν. Υπάρχουν εταιρείε οι οποίες συγκεντρώνουν δεδομένα, τα πακετάρουν και τα πουλάνε. Κατ' ουσίαν αυτό δεν είναι σκάνδαλο αλλά όσο υπάρχουν βέβαια όρια, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι γίνεται αυτή η συγκέντρωση δεδομένων εσείς εκπλήσεστε, εγώ πρέπει να σας πω όχι. Το 2008 η εκστρατεία του Ομπάμα ήταν πολύ προχωρημένη στο η μεμονωμένη στόχευση των ψηφοφόρων, αγόρασε δεδομένα από τους μεσάζοντες, τα συνδύασε με τους εκλογικούς καταλόγους, έκανε κάποιες συνεντεύξεις και μπόρεσε να εντοπίσει άτομα ως προς τι θα ψηφίσουν, τους αναποφάσεις τους επιπλέον Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε διαφορετικούς πελάτες με διαφορετική συμπεριφορά σε περίοδο εκλογών. Ε, αυτά είναι μεμονωμένα, ε, μονομένα άτομα τα οποία εντοπίστηκαν. Δεν είναι πολιτείες. Όλο αυτό γίνεται πολύ ενδιαφέρον γιατί τώρα βλέπουμε ότι αυτά επηρεάζουν τις εκλογές. Το 2016, μετά από 8 χρόνια, η εκστρατεία του Τραμπ, εδώ μια εταιρεία ισχυρίστηκε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ψυχογραφικά δεδομένα για άτομα για να προσθέσουν στο προφίλ των χρηστών έτσι ώστε να γίνονται ακόμα καλύτερες οι προβλέψεις. και τα βασικά στοιχεία που τόνιζαν ήταν ότι μπορούσαν να βρουν κατά πόσο ένα άτομο είναι ανοιχτό, ε, αν είναι ψυνείδητο, εξωστρεφές και διάφορα παρεμφερή, αν έχει νευρωτικές τάσεις, παρεμφερή. Πριν από κάποια χρόνια υπήρξε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Κάποιος έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αν δηλαδή δώσουμε στους ανθρώπους ένα ψυχολογικό ερωτηματολόγιο και πάρουμε απαντήσεις και το κάνουμε αυτό για ας πούμε 60.000 ανθρώπους, μπορούμε να βρούμε την ίδια άραγε απάντηση παρακάμπτοντας ε, το τεστ, δηλαδή χρησιμοποιώντας τη συμπεριφορά τους στην επιγραμμική online για να καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Και σκέφτηκαν να κάνουν αυτό το πείραμα. Δηλαδή άρχισαν να συγκεντρώνουν δεδομένα μέσα από το Facebook ε, και από άλλα app για να ε, φτιάξουν το προφίλ των ανθρώπων. Επίσης μπόρεσαν, πήραν άδεια για να αναλύσουν τα like που βάζουν και χρησιμοποίησαν αλγόριθμο για να μπορέσουν να κάνουν το συσχετισμό και κατέληξαν ότι πράγματι είναι δυνατόν να προβλεφτεί η προσωπικότητα χωρίς καν να γίνει αυτό το ψυχολογικό τεστ. Και βλέπετε εδώ αυτή τη μελέτη είναι περίπου 2-3 ετών πριν από δύο-τρία χρόνια, βλέπετε πόσο γρήγορα προχωρούν τα πράγματα. Από μία καθαρά ερευνητική μελέτη, μετά από τρία χρόνια, πάμε σε άλλη φάση και νομίζω ότι αυτό είναι μία πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιον κανονισμό. Το 2016, νομίζω το 2017, αυτή η ασφαλιστική εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποίησε τις ίδιες ψυχομετρικές πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αξιολογήσει ε, το, τη συμπεριφορά των οδηγών για να αξιολογήσει τον καθένα το τι θα πρέπει να πληρώνουν, να καταβάλουν ως ασφάλιστρα. Και πάλι λοιπόν χρειάστηκαν πολύ λίγα χρόνια για να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο προϊόν και σε μια συγκεκριμένη εκστρατεία. Νομίζω όλα αυτά ε, ήταν πολύ ενδιαφέροντα, αλλά δεν τελειώνει εκεί η ιστορία. Ε, Εν τω μεταξύ συνέβησαν και άρχισαν και άλλα πολλά πράγματα, ε, άρχισαν να εμφανίζονται αρνητικέ ειδήσει. Δεν στελιγάει και αυτό. Αυτό νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτοί οι δύο άνθρωποι στη φωτογραφία αποκλήθηκαν γορίλες από το Google από την ταξινόμηση της Google. Πριν από κάποια χρόνια δεν μπορούσε κανείς να κάνει αυτή την ταξινόμηση με βάση φωτογραφίες. Τώρα όμως γίνεται. Μπορεί κανείς ε, να εντοπίσει ένα άτομο, μια εικόνα. Ε, είναι μια τεράστια επιτυχία. Αυτοί είναι δύο Αφροαμερικανοί που χαρακτηρίστηκαν γορίλες. Αυτό ε, ήταν σκάνδαλο και τελικά ε, πολύ δυσάρεστο για την εταιρεία. Ζήτησαν ταπεινά συγγνώμη και τι έγινε, τίποτα. Ακριβώς αυτή είναι η εμπειρία μου, ότι δηλαδή λάθη γίνονται ε, σε καθημερινή βάση. Κανείς δεν το ήθελε αυτό, απλά ε, θα έπρεπε κανείς να ξέρει πώς συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα, πώς αξιολογήθηκαν, αν χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες ε, συνθήκες. Νομίζω ότι είναι <clears throat> φυσιολογικό να προκύπτουν και λάθη. Δηλαδή το σύστημα μαθαίνει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, ελαχιστοποιώντας τα λάθη. Αλλά όπως σας είπα, προέκυψε αυτό το σκάνδαλο. Και εδώ βλέπουμε ότι στις καταχωρήσεις της Google η Google έχει καταχωρήσει με βάση τις έρευνες που κάνει ο καθένας από εμά. Κάποιες σχέσεις έχουν με αφροαμερικανικά προϊόντα. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο και αυτό πάλι. Γιατί και πάλι το σύστημα ε, προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα κλικ, να οδηγήσει ανθρώπου ανθρώπους ε, στο να κλικάρουν. Άρα δηλαδή βρήκε κάποιο συσχετισμό ανάμεσα σε κάποια ονόματα και σε κάποια κλικ και αυτό ακριβώς όμως έπρεπε να κάνει το σύστημα. Το δυσάρεστο είναι ότι δεν μας αρέσει βέβαια στην κοινωνία μας να εφαρμόζουμε διακρίσεις έναν ε, των ανθρώπων. Αυτό βέβαια δεν το ξέρει το σύστημα και πάλι αν θέλετε στις γυναίκες. Ε, προβάλλονται περισσότερο πιο φτηνές εργασίες από ότι στους άντρες. Κανείς δεν θέλει να, είναι, ε, να επιβάλλει διακριτική μεταχείριση βάρος των γυναικών, απλά αυτό προκύπτει από το σύστημα με βάση τα δεδομένα και εάν ήδη υπάρχουν διακρίσεις στα data in the wild, αυτά όπως σας είπα τελικά οδηγούμε στο αποτέλεσμα. Η ε, μεγάλη ανακάλυψη θα ήταν να μπορέσουμε να κατανοήσουμε συγκαλυμμένες, συγκαλυμμένους συσχετισμούς για να είναι πιο σωστές οι προβλέψεις, αλλά ε, την διακριτική μεταχείριση και πώς θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα, αυτό προφανώς δεν γίνεται, άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα άλλο. Εγώ αναλύω δεδομένα εδώ και 12 χρόνια ε, και πρέπει να σας πω παίρνουμε χιλιάδες δεδομένα. Ε, έχουμε ε, πολλά βιβλία, 150 χρόνια υπάρχουν βιβλία στις αγγλικές βιβλιοθήκες και αυτά μπορούμε να τα αναλύσουμε. Υπάρχει δυστυχώς διακριτική μεταχείριση. Πρέπει όμως να το μάθουμε αυτό και πρέπει να κατανοήσουμε το τι θέλουμε να αποφύγουμε. Πότε κάτι μπορεί να είναι αποδεκτό, πότε όχι. Καταρχήν είναι θέμα κατανόησης. Η ιδέα να φτιάξουμε ένα μαύρο κουτί και αυτό να κάνει θαύματα και να μας προσφέρει χρήματα δωρεάν, αυτό νομίζω στην αρχή ήταν αφελές. Ε, ένα σύστημα που βασίζεται σε δεδομένα του παρελθόντος και που μπορεί να προβλέπει ποιος θα απελευθερωθεί με όρους, ε, ποιος θα επανέλθει, ποιος θα εξαφανιστεί, αυτό υπάρχει. Δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό, απλά λέω ότι ας ξεκινήσουμε από το να κάνουμε προβλέψεις, ξεκινώντας από κάτι απλό, αν ας πούμε θα αγοράσει κανείς γάλα αύριο ή όχι, να μάθουμε από αυτό και μετά να προχωρήσουμε. Αυτό συμβαίνει ήδη. Υπάρχουν διακρίσεις, κανείς ε, δεν είναι κακοπροαίρετος, αλλά αυτά συμβαίνουν. Όταν λοιπόν κάνουμε κάποιες προβλέψεις για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, νομίζω ότι είναι διαφορετικό το να κάνουμε προβλέψεις για ένα συγκεκριμένο άτομο. Γιατί οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα και κάποια πράγματα είναι απαράδεκτα. Εμείς λοιπόν ως ε, μηχανικοί ε, σε αυτό το τομέα είμαστε πολύ καλοί στο να ταξινομούμε δεξιότητες, να ταξινομούμε τους ανθρώπους, δυνατότητες πρόσβασή πρόσβασής τους, σε ευκαιρίες, ενημέρωση, σε μισθούς. Μην ξεχνάμε όμως ότι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα και η κοινωνία έχει ήδη οριοθετήσει ένα πλαίσιο για όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στις, ε, στα big data και στις ε, κατασκευασμένες ειδήσει ε, που συζητήθηκαν πολύ τον τελευταίο καιρό. Και πάλι, και αυτό έχει σχέση με την τεχνητή νομοθεσίνη, νοημοσύνη, γιατί το software προσπαθεί να δει που θα κλικάρατε, είναι το περίφημο filter bubble, το σύστημα λοιπόν με βάση όλα αυτά τα δεδομένα προσφέρει όλο και περισσότερα. Και αυτά ενδεχομένως να οδηγήσουν και σε πόλωση, γιατί επίσης είναι γνωστό ότι οι, οι σκέψεις μας επηρεάζονται από αυτά που διαβάζουμε ε, και αυτά που διαβάζουμε επηρεάζονται από τις απόψεις μας. Ε, άλλο ένα παράδειγμα, 160.000 ε, άνθρωποι εκτέθηκαν ε, στις ιστορίες του Τραμπ, ένας άλλος μεγάλος αριθμός εκτέθηκαν σε ιστορίες της Χίλαρη Κλίντον. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι εύκολο να καταλήξει κανείς το κατά πόσον μιλάμε για συγκεκριμένους εκλογείς στις ΗΠΑ. Αυτή η όλη ιδέα πίσω από αυτά είναι ότι έχουμε το μηχάνημα μάθησης προ τα δεδομένα, συν τα προσωπικά δεδομένα, που καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αν όμω υπάρχει κάποια προκατάληψη, ε, το σύστημα το εντοπίζει και μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Πού ε, φτάνουμε λοιπόν. Φτάνουμε στο εξή. Αυτό που έχουμε κατασκευάσει είναι ένα νέο μέσο μεσο ενημέρωση, με την έννοια του Μάρσαλ Μακλούαν είναι ένα νέο μέσο. Δεν είναι όπως το τηλεγράφημα ή το τηλέφωνο ή η τηλεόραση. Δεν είναι ε, ένας ε, αγωγός που μεταφέρει παλμούς ε, μπορεί να αποφασίσει το τι θα δείτε, τι πρέπει να συστηθεί είναι ένας ε, πολύ καλός ε, λόγος ε, και ένα πολύ καλό μέσο γιατί θυμάται τα πάντα. Αυτά έγιναν το 2017. Αυτά είναι ότι έχουμε ένα νέο μέσο μαζικής ενημέρωσης που είναι τελείως διαφορετικό από αυτά που είχαμε κατά το παρελθόν. δεν είναι σκευωρία, δεν έχουμε hackers από τη Ρωσία, έχουμε ένα νέο μέσο και διαπιστώσαμε όμως ότι πλέον δεν είναι όλα τέλεια, περί αυτού πρόκειται. Η ιδιωτική σφαίρα μας απασχολεί, μας ανησυχεί, οι προκαταλήψεις, οι διαφάνειες, ε, η μετατόπιση εξουσίας, αλλά όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι η τεχνητή νομοσύνη είναι καταδικαστέα. Εγώ θα συνεχίσω να ασχολούμαι με την τεχνητή νομοσύνη στο πλαίσιο των ε, σωστών κανονισμών. Υπάρχει λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη και οι μηχανές μάθησης ε, για διάφορους λόγους. Εμείς μπορούμε να υποφεληθούμε από όλα αυτά. Ας δούμε τώρα λιγάκι αυτό. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα νέο μέσο και το βάλαμε αυτό στο κέντρο της ζωής μας την πρώτη φορά που έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη από την οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Μπορεί να μας επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη, μας κοιτάει, μαθαίνει από εμάς, μπορεί να μάθει για μας πράγματα που δεν μας αρέσουν. Ε, αυτό δεν μπορούμε, πρέπει να το δεχτούμε ε, και δεν μπορούμε να την αποφύγουμε την τεχνητή νοημοσύνη η ε, υπόσχεση στην αρχή ήταν σχετικά με τους ενδιάμεσους, ήταν πολύ αισιόδοξη. Βασικά αυτούς τους αντικαταστήσαμε με αλγόριθμους, τους ενδιάμεσους. Νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντική θέση. Οι αλγόριθμοι πλέον βρίσκονται στην ίδια θέση που ήταν παλαιότερα οι ενδιάμεσοι. Εκείνοι αποφασίζουν τι πληροφορίες θα δοθούν στους ανθρώπους. Και έτσι φτάνουμε σε μια νέα σημαντική πρόκληση για όλους μας, που είναι και το θέμα της μενής συνάντησης, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε με τις ευφυείς μηχανές. Αν δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε, υπάρχουν και ε, είναι προκλητικές, πώς μπορούμε να συνεπάρξουμε. Αυτό είναι το θέμα κατ' ουσίαν, το οδηγό νήμα της ομιλίας μου. Πώς μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες ότι θα υπάρχει δικαιοσύνη, ε, διαφάνεια, λογοδοσία, πώς μπορούμε να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά τι μπορεί να είναι αποδεκτό και τι όχι. Δεν θέλουμε να κλείσουμε την τεχνητή νομοσύνη, θέλουμε μόνο να μην προκαλεί ζημιά σε κανένα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το γενικό πλαίσιο ε, κανόνων είναι πολύ καλό, όσο το διαβάζω μου και καλύτερα, δεν λύνει τα πάντα, αλλά λύνει κάποια θέματα Πρέπει όλα αυτά να τα πάρουμε σοβαρά υπόψη μας. Και ένα πράγμα που θέλω να συστήσω στο Κοινοβούλιο είναι το εξής. Δέστε πώς θα εφαρμόσετε αυτόν τον κανονισμό. Εάν ε, αναγκαστείτε να αποκηρύξετε ορισμένα πράγματα για να υιοθετήσετε μια ε, νέα συσκευή, αυτό δεν είναι σωστό εάν οι άνθρωποι σας πούν ότι δεν μπορούμε πια να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νομοσύνη με τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να απαντήσει κανείς ότι ακριβώς γι' αυτό ας συζητήσουμε γιατί όλα αυτά μπορούν να γίνουν με ένα σχετικά διαφορετικό τρόπο. Θα κλείσω, τελειώνω. Το θέμα είναι ότι στο μέλλον θα συγκεντρώνονται περισσότερα δεδομένα γιατί Έχουμε μια κοινωνία που θα χρησιμοποιεί μόνο πιστοτικές ε, κάρτες. Ορισμένοι συναδελφοί μου ε, έχουν ενθουσιαστεί πάρα πολύ ε, σχετικά με τους αλγόριθμους και τους κανονισμούς, σχετικά με τους αλγόριθμους, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτή, αυτό το μη γραμμικό feedback θα πρέπει να μας καθιστά επιφυλακτικούς. Υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί σχετικά με την κοινωνία που δεν χρησιμοποιεί ε, ρευστά διαθέσιμα. Κάτι πρέπει να κάνουμε και ταχύτατα. Θα ακούσετε ότι αν όμως δεν υπάρξουν κανονισμοί, αυτό θα είναι εις βάρος της οικονομίας. Αλλά να έχετε κατά νου ότι ακόμα υπάρχει αρκετός χρόνος για να προγραμματίσουμε. Και συγκεκριμένα αυτές οι τρεις έννοιες, αλγοριθμική, κανονισμοί, κοινωνία χωρίς ε, νομίσματα, αυτό και πάλι σημαίνει ότι έχουμε ενδιάμεσους. Ενδιάμεση ποιοι είναι, είναι οι αλγόριθμοι. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και θέλω να κλείσω με μια αισιόδοξη νότα. Γιατί νομίζω ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε σωστά. Και πώ θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη, αυτό ε, εναπόκειται σε εμά. Νομίζω ότι μπορούμε να, κατα... εξηγήσουμε καλύτερα την τεχνητή νοημοσύνη, ίσω να χρειαστούμε νέου θεσμού. Οι άνθρωποι μιλάνε ε, πάρα πολύ για ε, την ε, πιστοποίηση την πιστοποίηση με βάση τους αλγόριθμους. Νομίζω ότι πρέπει να διερωτηθούμε. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη σε δημόσιους χώρους. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, δεν είναι ότι θέλω να αναχαιτήσω τίποτα. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και παρεπιπτόντως όλοι μας έχουμε πληρώσει, όλοι μας έχουμε καταβάλει χρήματα, είναι δημόσιο το χρήμα, ε, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, χρειαζόμαστε τους σωστούς νόμους, ε, τα σωστά βήματα, πολιτισμικά βήματα και ε, νομίζω ότι τελικά θα επεκταθεί όλο και περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη. Το 17 δεν ήταν εξαίρεση, είναι η πρώτη χρονιά, θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα παρεμφερή. Αυτά να μην τα ξεχνάμε, να τα έχουμε πάντα κατά νου. Χρειαζόμαστε περισσότερες ιδέες. Η βασική ιδέα είναι σημαντική. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Όλα αυτά είναι οι παρενέργειες, αν θέλετε, τα παρελκόμενα περισσότερο ε, αυτών των θετικών που έχουν προηγηθεί. Εναπόκειται λοιπόν σε εμά, όπως σας είπα, το να έχουμε κατά νου το μέλλον μας. Δεν είναι θέμα των μηχανικών του κλάδου, ε, δεν πρόκειται, για αυτούς, ε, δεν πρόκειται καν για αυτούς κάποιες λύσεις είναι τεχνικές. Ε, πρόσφατα οι ιδέες είχαν προκύψει από φιλοσόφους, καλλιτέχνες, ε, επιχειρηματίες. Το θέμα είναι να προσθέσουμε πάρα πολλές καινούργιες ιδέες σε αυτή τη συζήτηση. Και ευχαριστώ πολύ που μας, με προσκαλέσετε. Ας περάσουμε τώρα στην πρακτική εργασία. So besides being engineer, you're a politician, you have to ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ, καθηγητή, για αυτή την θαυμάσια παρουσίαση. Έχω κάποιες ανησυχίες, αλλά μου απαντήθηκαν και κάποια ερωτήματα. Σίγουρα θα πρέπει να οργανώσουν περισσότερες τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί ο τομέας είναι τεράστιος, άπειρος και μόλις ξεκινάμε. Θα περάσω τώρα το λόγο στους πανελίστες μας θα υπάρχει και χρόνο στο τέλος των παρουσιάσεων να υποβληθούν ερωτήσεις και να δοθούν απαντήσεις. Ο David Wildon είναι διευθυντής στο Sky και θα είναι ο επικεφαλής του επόμενου πάνελ. Κάνει, ανήκει σε μια ομάδα που κάνει πολιτική ανάλυση. Τον συνάντησα στην, πριν γίνει το Brexit προσπαθούσαμε να συζητήσουμε και να καταλάβουμε πού πήγαινε το πράγμα. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα μιας απόφασης ε, κλινικής ε, ε, αναμέτρησης ενός δημοψηφίσματος κτλ. Έχετε το λόγο κύριε David Wildon για να καλέσετε τους πανελίστες από το MIT, από το Elsevier, από το Πανεπιστήμιο του Sheffield, το Google, την Google και το Facebook. Ε, ελάτε, ελάτε όλοι παρακαλώ στο βήμα. And we have translation, uh, French, Γαλλικά, Ισπανικά και Ελληνικά. Ε, είναι οι γλώσσες οι οποίες ε, μεταφράζονται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας, εάν θέλετε να ακούσετε τη διερμηνία. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ήταν ε, εντυπωσιακή η παρέμβαση που ακούσαμε. Η μόνη πολιτική πρόβλεψη που πέτυχα ήταν αυτή για τον Brexit. Όχι γιατί έκανα καμιά ιδιαίτερα περίεργη ανάλυση με φοβερούς αλγορίθμους, είναι απλώς γιατί έφυγα και ταξίδεψε μακριά από το Λονδίνο μερικέ φορές. Μόνο αυτό χρειάστηκε. Όλοι είμαστε μέσα στη φούσκα μας, μέσα εκεί ζούμε. Ε, με εντυπωσίασε αυτή η συζήτηση που ξεκινήσαμε, γιατί πραγματικά είχα την αίσθηση ότι κάποιο μου δίνει νέε ιδέες και ότι σπάμε κάτι μπαγιάτικο, παλιό, ξεπερασμένο που κάνουν οι πολιτικοί με τον κλάδο. Και τώρα λοιπόν θα έχουμε αυτό το πάνελ συζήτησης ελεύθερα θα ήθελα να μιλήσουμε. Θα ήθελα ο καθένας να μιλήσει για 10-15 λεπτά και εν συνεχεία θα του θέσουμε ερωτήσει. από το κοινό. Θα ξεκινήσουμε με τον Μίχαελ Μπλέτσα που έχει μία 20χρονη καριέρα στο εργαστήριο για τα ΜΜΕ ε, του MIT. Είναι πληροφορικάριος Μάλιστα έχει δημιουργήσει και ένα κομπιούτερ για παιδιά. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό επίτευγμα στο βιογραφικό του. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν τη δική του άποψη καταρχήν, του κύριου Μπλέτσα. Θέλω να επαναλάβω κάποια από τα πράγματα που ακούσαμε από τον προηγούμενο μιλητή από μια διαφορετική οπτική σκοπιά. Ακούσαμε την άποψη του μηχανικού. Αλλά θα ήθελα να κάνω και κάποιες υπεραπλουστεύσεις, κάποιες σχηματοποίησεις, ούτως ώστε να περάσει το μήνυμα ε, πολύ πιο άμεσα, αν θέλετε. Πρώτο ερώτημα για την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι, είναι πραγματική επανάσταση, είναι η επαρχία της επανάστασης ή είμαστε στο τέλος της επανάστασης. Η βασική ιδέα για την τεχνητή νοημοσύνη, τα βασικά μαθηματικά υπάρχουν τουλάχιστον από το 1986 και αυτό που σήμερα χρησιμοποιούμε για την εκμάθηση της μηχανής είναι ε, νευρονικά δίκτυα και το deep learning, βαθιά ε, μάθηση. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα νευρονικό δίκτυο με πολλά στρώματα, που αυτά ε, τα επινοήσαμε στη δεκαετία του 50 και του 60. Είμαι σε λιγάκι περίεργη θέση εδώ, γιατί ε, είμαι μαθητής του κυρίου Μίνσκι, και τώρα μιλάω για το machine learning, για την εκμάθηση μηχανής στον 21ο αιώνα. Το 1969 μιλάμε ε, για δύο ανθρώπους οι οποίοι δημοσίευσαν ένα βιβλίο στο MIT και μιλήσαν για θεωρητικές απομιμήσεις νευρονικών δικτύων και πολλοί τους κατηγόρησαν ότι στην πραγματικότητα πέταξαν αυτή την έρευνα, τη φήμωσαν, τη σταμάτησαν. Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια ε, τόσο ώστε ο Τζέφρι Χίντον από το Πανεπιστήμιο του Τορόντου να φτιάξει έναν αλγόριθμο για να εκπαιδεύσει αυτά τα νευρονικά δίκτυα. Ο, προφέσορ, ο καθηγητής αυτός ε, επινόησε αυτόν τον αλγόριθμο. Δεν ήταν πολύ πρακτικός γιατί δεν υπήρχαν πολλοί πόροι και πολλά δεδομένα εκμάθησης εκείνη την εποχή. Χρειάστηκαν λοιπόν κάποιες δεκαετίες και χρειάστηκε η μεγάλη πλατφόρμα του ίντερνετ για να δώσει αυτά τα πολλά ε, ε, δεδομένα και χρειάστηκαν κάποιες ε, υπολογιστικές δυνατότητες. Η βασική αρχιτεκτονική για τα δίκτυα αυτά είναι αυτά που χρησιμοποιούμε, μπορούσαμε για παιχνίδια υπολογιστή και για γραφικές παραστάσεις. Άλλη ηρωνία εδώ πέρα. Αλλά φτάσαμε εκεί που φτάσαμε σήμερα. παντού βρίσκουμε την τεχνική νοημοσύνη μπροστά μας. είναι εντυπωσιακό το πόσες πολλές εφαρμογές έχει και πώ πολλές εφαρμογέ τη χρησιμοποιούν. Αν ε, λάβουμε υπόψη μας όλες οι υπόλοιπες εφαρμογές, ε, υπάρχει μία που είναι πολύ πιο σημαντική από όλες μαζί. Δηλαδή, ε, η στόχευση κάποιων διαφημίσεων σε συγκεκριμένους χρήστες του ίντερνετ. Από εκεί βγαίνουν τα λεφτά. Και έχει όμως και κάποια, κάποιες παρενέργειες. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι είμαστε στο τέλος μιας τεχνολογικής επανάστασης και όπως συμβαίνει με κάθε επανάσταση, τώρα θα πρέπει να ξαναδούμε πού βρισκόμαστε, ε, να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ας πούμε και να τα ανασυνθέσουμε. Ένα άλλο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, για το οποίο έχει γίνει πολλής λόγος, είναι ότι ως συνήθως η τεχνολογία ε, Ήτανε πρώτα και μετά η επιστήμη. Ξέρουμε τα φτιάχνουμε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργούν. Είναι σαν μαύρα κουτιά. Για πολλούς ανθρώπους. Για τους περισσότερους θα έλεγα. Ένα απλό παράδειγμα που αναφέρθηκε και πριν. Δεν ξέρω πόσοι ε, έχετε ακούσει για το AlphaGo και το AlphaGo 0, 0. Είναι νευρονικά δίκτυα της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιήθηκαν για να ε, παίξουμε το παιχνίδι του Go, αυτό το παιχνίδι που λέγεται Go, που θεωρείται πολύ πιο δύσκολο ε, σε σχέση με το σκάκι, ε, γιατί έχει πολύ περισσότερες κινήσεις. Στην πρώτη εκδοχή του AlphaGo χρησιμοποιήθηκαν παιχνίδια, υπάρχοντα παιχνίδια που τα έχουμε παίξει, για να εκπαιδεύσουμε τα νευρονικά αυτά δίκτυα και φυσικά νίκησε πολύ εύκολα το μηχάνημα τους ανθρώπου, ανθρώπους, τους Και μετά χρησιμοποίησα μια άλλη δέκα. Αντί να χρησιμοποιήσουμε πραγματικά παιχνίδια, θα δώσουμε τους κανόνες. Και να παίξεις εναντίον του Μπορείς να παίξει ε, εναντίον του εαυτού για να μάθεις. Έμαθε το μηχάνημα πολύ καλά. Νίκησε τις προηγούμενες εκδοχές του παιχνιδιού και φυσικά όλους τους ανθρώπινους πρωταθλητές. και μάλιστα ε, τις κινήσεις που κάνει δεν μπορούμε να τις εκφράσουμε σε μαθηματικά απόλυτα. Αυτό το σημείο πρέπει να το κρατήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν γνωστό από την αρχή. Δηλαδή, προσπαθούμε να θεωρήσουμε την... Ε, προσπαθούμε να θεωρήσουμε ότι η νοημοσύνη είναι κάτι που μπορούμε να το εξηγήσουμε. Υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη εδώ και πολλά χρόνια. Κάνας ε, δεν θεωρεί, ας πούμε, ότι το να παίζει κανεί σκάκι με το μηχάνημα είναι τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί λίγα, λίγο πολύ του καταλαβαίνουμε του αλγόριθμου. Ε, το ίδιο ισχύει και με τα συστήματα, διάφορα συστήματα που υπήρχαν στο παρελθόν, συμβολικά σύστημα κτλ. Ε, με την ε, μηχανή μάθηση είναι πιο περίπλοκο. δεν μπορούμε να το καταλάβουμε κάτω μαθηματικά το πώς λειτουργεί. Σίγουρα όμως ε, θα προχωρήσουμε πολύ περισσότερο από εδώ που είμαστε σήμερα. Ε, η επιστήμη θα ακολουθήσει την τεχνολογία, αλλά αυτό μας φοβίζει. Το τρίτο σημείο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι φυσικά ε, επειδή έχουμε κάτι μπροστά μας που δεν το καταλαβαίνουμε απόλυτα, μας φοβίζει. Κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα προέκυψε χωρίς να το θέλουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη, ε, η εκμάθηση, η, μηχανή μάθησης προέκυψε κατά τύχη. Και εξού και οι φόβοι μας. Καθώς θα προχωρούμε, σε ό,τι αφορά τη διάδοση ας πούμε ειδήσεων, ο κύριος ε, Χριστιανίνη το εξήγησε πάρα πολύ καλά το θέμα. Στην πραγματικότητα αντικαταστήσαμε τους δημοσιογράφους με αυτά τα συστήματα, με αυτά τα φίλτρα της τεχνητής νοημοσύνης και η αντικατάσταση αυτή δεν πήγε πολύ καλά, δεν λειτουργήσε πολύ καλά. Αυτό φαίνεται προς το παρόν. Ε, μπορούμε να το διορθώσουμε, φυσικά μπορούμε. Θα το διορθώσουμε χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, όμως όχι. Όχι με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν διορθώνεται το πράγμα. Μην ξεχνάτε ότι τελικά η σημερινή τεχνητή νοημοσύνη κάνει το εξή πράγμα πολύ καλά. Ε, συνδυάζει κάποια στοιχεία που τροφοδοτούμε στο μηχάνημα και δίνει κάποια αποτελέσματα. Αυτό κάνει. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η δεξιότητα, αλλά είναι πολύ περιορισμένη. Εγώ είμαι κάποιος που πιστεύει ότι τελικά θα υπάρξει τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα κάνει παραπάνω, πράγματα. Θα διαβάζει, α πούμε. Όμω η σημερινή τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ στενή νοημοσύνη. Όταν φτάσουμε σε μια γενικευμένη νοημοσύνη, δεν αρκεί απλώ να προσθέσουμε πολλές ε, μορφές στενής τεχνητής ε, νοημοσύνη για να φτάσουμε σε κάτι γενικευμένο, σε μια γενική ε, νοημοσύνη. Θα πρέπει να ξαναπάμε πίσω στα νευρονικά δίκτυα, να καταλάβουμε επίση ε, να μας βοηθήσει η επιστήμη, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η ανθρώπινη νοημοσύνη για να υπάρξει μια επανάσταση. Πάντως, η σημερινή τεχνητή νοημοσύνη θα γίνεται όλο και πιο χρήσιμη, θα γίνεται όλο και πιο τέλεια. Δεν θα πρέπει στην πραγματικότητα όμως να μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε για κομπιούτερ που βοηθούν τους ανθρώπους. Υπήρξαν παρενέργειες, ανεπιθύμητες ε, ενέργειες και δεν νομίζω ότι η λύση είναι να πούμε ότι αυτός κάνει να δουλεύει στον τομέα της τεχνικής, ε, τεχνητής νοημοσύνης και αυτός όχι. Χρειαζόμαστε επιστήμονες από, όλες τις, ε, από όλους τους κλάδους. Το, αυτό που με φοβίζει προς το παρόν δεν είναι ότι θα ξεφύγει η τεχνητή νοημοσύνη και θα κάνει ό,τι θέλει ας πούμε, αλλά φοβάμαι ε, τους ε, αδαείς ηγέτες οι οποίοι δεν σκέφτονται τις συνέπειες της τεχνολογίας που δίνουν στον κόσμο. Δεν φοβούμε αυτή τη στιγμή δηλαδή τις μηχανές οι οποίες θα παίρνουν αποφάσεις για λογαριασμό μας. Και εδώ θα ήθελα να σταματήσω. Ευχαριστώ. Θα έπρεπε από την αρχή να σας πω ότι ένα ρόλο που θέλω να παίξω είναι ε, να ε, κάνω εγώ ερωτήσει ε, που δεν θέλετε ίσω να κάνετε εσείς. Θα προσπαθήσω να τον παίξω καλά αυτό το ρόλο. Μιχάλη, ένα πράγμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ένα πράγμα που έχω διαβάσει εδώ. Είσαι ένα επαείων της τεχνολογίας, ο οποίο κατ' ουσίαν πρέπει να τοποθετήσω εξή. Διαφάνεια χρησιμοποιήθηκε ως λέξη. Αλλά έχω μια ερώτηση. Αν τελικά οι εταιρείε οι τεχνολογικές που δουλεύουν σε αυτό το χώρο ήταν πιο διαφανείς, αν πρόκειται να δημοσιεύσουν τους αλγορίθμους τους για να μπορούμε να τους μελετήσουμε, άνθρωποι σαν και σένα θα μαθαίνανε από αυτούς τους αλγορίθμους. Είναι απλό δηλαδή να γίνει αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι απλό. Προφανώς δεν είναι απλό. Η διαφάνεια μόνη τη από μόνη τη, ε, δεν επιλύει τίποτα, εκτός αν έχουμε ανθρώπους που καταλαβαίνουν περί τίνο πρόκειται. Και νομίζω σε αυτή την περίπτωση το περιεχόμενο των αλγορίθμων είναι σημαντικότερο γιατί έχουμε να κάνουμε με περίπλοκες ιδέες ε, το να λέμε ή να πιστεύουμε ότι όλοι θα τα καταλάβουν όλα αυτό είναι τοπικό δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύει Πρέπει όμως να γνωρίζουμε το στόχο. Και επίσης πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί ε, που αφορούν στο μέγεθος ε, της ε, συγκέντρωσης και στην πυκνότητα της συγκέντρωσης των ενδομένων. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε, να περιορίσουμε τις ανεπιθύμητες συνέπειες και προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε τις θετικές προεκτάσεις. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κόλμαν, ο οποίος είναι ε, πρόεδρος ε, την, ε, ε, ε της Διεθνούς Ένωσης Εκδοτών. Ε, ο Μιχάλης, ο Μιχάλης Κόλμαν, μάλλον ο Μιχάλης ήταν είχε σχέση με τους υπολογιστέ, τώρα πάμε σε αστροφυσικό. Ακριβώς το αντίθετο. Ε, επιτρέψτε μου λοιπόν να ε, απευθυνθώ με μεγάλη μου χαρά σε επιστήμονες, σε συναδέλφους. Από τότε λοιπόν πριν από 30 χρόνια εμφανίστηκε ε, το δίκτυο, το διαδίκτυο. Υπήρξαν εξελίξεις που επηρεάζουν τη ζωή μας. Ε, η Apple, η Microsoft, η Amazon εμφανίστηκαν αυτά τα ονόματα που είναι από τα πιο αναγνωρισμένα στον κόσμο και τώρα πια είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες. Η Google μας βοηθάει να ε, βρούμε τις απαντήσεις, μπορούμε να βρούμε βίντεο στο YouTube και όλα αυτά ε, μπορούμε επίσης να τα βρούμε και στην Amazon και στην Microsoft. Μπορούμε να τα κάνουμε πάρα πολύ εύκολα. Αυτές λοιπόν οι εταιρείε ε, άλλαξαν τη ζωή μας. Παράλληλα, πάρα πολλοί διορωτώνται ε, ποιε είναι οι επιπτώσεις, τι μπορούν να καταφέρουν αυτές οι λίγες εταιρείε στις κοινωνίες που να είναι τόσο σημαντικό. Πριν από λίγες εβδομάδες δημοσιεύτηκαν σχόλια από το Facebook και νομίζω για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι πλέον γνωστό ότι τα αποτελέσματα ή αναζητήσεις μέσω της Google μπορούν να ε, υποστούν δόλιους ε, χειρισμούς ε, για συγκεκριμένους σκοπούς. Ε, βασικά το να διαδώσει κανείς ε, καλές πληροφορίες είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια με τον τρόπο αυτό οι κακές πληροφορίες ε, είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές και αυτές οι πληροφορίες μας κατακλείζουν. Μερικοί βλέπουν ότι οι υπηρεσίες που εξερτώνται από κλικ, οι πληροφορίες αυτές ίσως να είναι σημαντικές. Θα ήθελα όμως να πω ότι οι η τεχνολογικοί κολοσσοί φέρουν ευθύνη, ίσως ε, θα πρέπει να βρουν κάποια νέα μορφή έμπνευση. Ας δούμε τώρα τι γίνεται με τους εκδότες. Οι εκδότες έχουν να τερματίσουν σημαντικό ρόλο στο να αναχαιτήσουν την περαιτέρω διάδοση των κατασκευασμένων ειδήσεων. Τα τελευταία 20 χρόνια όλο και περισσότερο μετακινηθήκαμε προς online πλατφόρμες όπως και οι εταιρείε οι τεχνολογικές. Εγώ ε, έχω μια συγκεκριμένη εμπειρία από την Elsevier και μπορούμε να σε εγγυηθούμε ότι το υλικό που ε, παράγουμε εμείς ε, πληρεί τους κανόνες, ε, έχει ελεγχθεί, συνταχθεί, ελεγχθεί, μετά έχει αναθεωρηθεί και πάλι αναθεωρηθεί για να βελτιωθεί περαιτέρω ποιότητα. Και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι υπάρχει σωστή επιμέλεια έτσι ώστε το υλικό αυτό να παραμένει προσπελάσιμο και στο μέλλον. Με άλλα λόγια, εμείς αναλάβουμε την ευθύνη του περιεχομένου που δημοσιεύουμε. Σημαίνει άρα γι' αυτό ότι η δουλειά μας είναι τέλεια σε τελική ανάλυση και οι εκδότες είναι εταιρείε ε, όπως ε, και άλλοι ομολογοί μας και αυτοί είναι άνθρωποι. Μετά λοιπόν από έρευνες ε, μπορεί να περάσει, να ξεφύγει και ένα άρθρο που δεν θα έπρεπε. Ευτυχώς όμως υπάρχουν αυστηρές διαδικασίες για να αντιμετωπίζονται αυτές τέτοιου του άρθρα και να διορθώνονται. Βλέπουμε επίσης ε, ότι οι εκδότες ε, προσχωρούν στην τεχνολογία σήμερα. Βέβαια η ψηφιακή τεχνολογία όχι μόνο κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας, αλλά βελτιώνει και το περιεχόμενο που δημοσιεύει. Το διαδίκτυο ήταν ένα άλμα προς τα εμπρός, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο, να μπορούμε να το διαμορφώσουμε. Και τα τελευταία χρόνια με την τεχνολογία εξόριξης δεδομένων, με τις μηχανές μάθησης, μπορούμε επιπλέον να επεξαργαζόμαστε το περιεχόμενο και με άλλους τρόπους. Όχι μόνο να το διαβάζουμε, να το αφομοιώνουμε και διαφορετικά. Οι ε, εκδότες προσφέρουν κάποια επιλογή και ο αναγνώστης, χρησιμοποιώντας τη δική του τη λογική, προσπαθεί να αποκτήσει γνώση μέσα από αυτά τα δεδομένα. Η ε, τεχνητή νομοσύνη μας δίνει τη δυνατότητα να αποκομίζουμε γνώση και με συγκεκριμένα γραφήματα. Αλλά ε, εμείς χρησιμοποιούμε τις μηχανές μάθησης και την τεχνητή νομοθεσίνη με αυστηρούς ε, όρους. Θα αναφέρω και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Ε, μπορούμε να έχουμε ιατρικές γνώσεις με εύπεπτα λεπτό τρόπο μπορεί κανείς πάρα πολύ εύκολα να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για να μπορεί να λάβει αποφάσεις υποποίηση. Και με τον τρόπο αυτό ενδεχομένως σώζονται και ζωές. Ε, γιατί οι κακές πληροφορίες ε, είναι καθοριστική σημασίας για, την, ε, για να σωθεί μια ζωή οι εκδότες μπορούν να εγγυηθούν ότι το περιεχόμενο που έχουν στα χέρια τους όχι μόνο είναι αξιόπιστο αλλά και αποτελεσματικό. Οι εκδότες λοιπόν χρησιμοποιούν την τεχνολογία εξόριξης δεδομένων και τους αλγόριθμους για να έχουν πιο ακριβή δεδομένα. Ε, επίσης συνδυάζουν τη τεχνολογία με την ανθρώπινη ευθεία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτές οι εξελίξεις δεν μπορούν να είναι εις βάρος της ποιότητας. Η εμπιστοσύνη προς εμάς ε, είναι κάτι που μας απασχολεί και θα συνεχίσει να μας απασχολεί και στο μέλλον. Και εφόσον μιλάμε για την εμπιστοσύνη υπάρχουν πολλά θέματα που μας ανησυχούν τα τελευταία χρόνια. Οι εκδότες όλο και περισσότερο διαθέτουν κάποιο περιεχόμενο ε, μέσα από πλατφόρμες ε, και πριν τυπωθούν συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτή η μετατόπιση έχει μια σκοτεινή πλευρά. Ανησυχούμε πάρα πολύ σχετικά με επιστημονικά δεδομένα τα οποία δεν έχουν φτάσει στην τελική τους φάση, δηλαδή δεν έχουν ελεγχθεί ποιοτικά. Ε, όσον αφορά τις ιατρικές ε, πληροφορίες που και αυτές ανεβαίνουν στο διαδίκτυο. Ένα άρθρο χωρίς να έχει αξιολογηθεί ως προς την ποιότητά του, αυτό υπάρχει. Εμείς όλο και περισσότερο βασιζόμαστε στους αλγόριθμους. Θα έπρεπε όμως να υπάρξει και αξιολόγηση αυτών των αλγορίθμων με βάση αυτά που ακούσαμε. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερο επίπεδο διαφάνειας ε, σχετικά με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Εάν μας ενδιαφέρει πραγματικά το περιεχόμενο, περιεχόμενο που δημοσιεύουμε θα έπρεπε οι εκδότες να, να προχωρούν πολύ προσεκτικά. Στις αρχές αυτού του έτους η Elsevier ως μια εταιρεία Big Data ε, εμείς απευθυντήκαμε σε διάφορες οργανώσεις του κόσμου ε, για να δούμε τα δικά του αποτελέσματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές λοιπόν οι πληροφορίες, αυτές τις συγκεντρώσαμε ε, και βλέπετε εδώ ε, τις επικεφαλίδες ε, που πραγματικά σοκάρισαν τους Ιάπωνες. Ε, βλέπουμε το τι αποκαλύφθηκε μέσα από πολύ καθαρά επιστημονικά άρθρα. Και αυτό που βλέπουμε εδώ, πάνω πάνω κιόλας, είναι ότι έχουμε τις Αμερικανικές εταιρείες, τη Microsoft, τη Google που κυριαρχούν στον κλάδο. Υπάρχει και ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, η RNS, που έχουμε και Γάλλους συναδέλφους εδώ από αυτή την εταιρεία. Έχουμε έχουμε και ισχυρή εκπροσώπηση από την Ασία και από την Κίνα. Ε, στους 100 έχουμε μόνο μία Ιαπωνέζικη εταιρεία, έναν φορέα και αυτό ήταν ε, ένα σοκ για τους Ιάπωνες. Ας δούμε τι γίνεται με τους ε, Ευρωπαίους. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Βλέπουμε λοιπόν στις, στους πρώτους 25, στις πρώτες 25 εταιρείε είναι οι γαλλικές Σακλέιν Χαϊά και μετά όπως βλέπετε στις πρώτες 25 είναι Imperial, Oxford. Δεν εκπλήσει το ότι ε, έχουμε τους ε, συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο ασχολείται πάρα πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε επίσης να ισχυριστούμε ότι η Ευρώπη ε, είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με τις ΗΠΑ και την Ασία όσον αφορά την τεχνητή νομοθεσία. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι τεχνολογικές εταιρείε είναι όλο και περισσότερο σαν τους εκδότες. Παρουσιάζουν ένα περιεχόμενο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι εκδότες σιγά σιγά μετατρέπονται σε τεχνολογικές εταιρείε, βασίζονται στην εξόριξη δεδομένου και στην τεχνητή νομοσύνη για να μπορέσουν να έχουν πληροφορίε από ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο φαινόμενο. Εμείς ε, και οι εκδότες και οι εταιρείε είμαστε υβριδιακοί οργανισμοί, έχουμε θεματολόγιο με πολλούς ε, στόχους. Αν λοιπόν θέλουμε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την ανθρωπότητα θα πρέπει να εξισορροπούμε το περιεχόμενο και την τεχνολογία σε σχέση με όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στους εκδότες και τις εταιρείε, τις τεχνολογικές για να μπορούμε να έχουμε ισορροπίες και έλεγχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εσείς και εγώ προερχόμαστε από τον παλιό κόσμο των ΜΜΕ. Ε, χρησιμοποιείται ανθρώπους για να ελέγξουν τα επιστημονικά έγγραφα. Εμείς χρησιμοποιούμε εκατοντάδες ε, δημοσιογράφους ε, σε όλη την Ευρώπη για τα κανάλια μας και χρησιμοποιούμε ε, τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο και να προωθήσουμε την επιχείρηση ας πούμε, της, στην οποία ανήκουμε και να κάνουμε και τον έλεγχο. Οι ε, επιστήμονες στην περίπτωσή σας ας πούμε, κάνουν με αυτόν τον τρόπο πιο παραγωγική δουλειά. Μία ερώτηση για το δικό σας κόσμο και την τεχνητή νοημοσύνη. Ε, ασχολείστε με περίπλοκα θέματα, με θέματα που είναι ζωτικής σημασίας για την ζωή των ανθρώπων, ειδικά στον τομέα της υγείας και της ιατρικής αν έχουμε την απόλυτη διαφάνεια, πώς είναι δυνατόν σε ένα κόσμο τεχνητής δοημοσύνης που μαθαίνουν οι μηχανές να έχουμε ε, προσωπική και ηθική λογοδοσία. Θα είναι ποτέ αυτό δυνατόν? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα πρέπει να απαντήσει πολιτικό και όχι εγώ. Αλλά μην ξεχνάτε ότι όταν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία τεχνητή νοημοσύνη, ε, μιλάμε για περιεχόμενο που έχει ήδη επιμεληθεί ε, και φροντιστεί. Ε, ας πούμε, μπορούμε να έχουμε βιβλία από γιατρούς, ε, paper από ε, επιστήμονες και όταν χρησιμοποιείτε την τεχνητή την τεχνητή νοημοσύνη εκεί, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ υψηλή ποιότητα. και θα πρέπει να υπάρχει ας πούμε, και ένα στοιχείο ε, διοντολογία, ηθικό εκεί μέσα. Ε, ένα άλλο ε, ο Ανδρέας Βλάχο από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλ. Ο Ανδρέας, είναι πολύτιμος εδώ με αυτά που ξέρει, γιατί είναι ένας από τους ε, βασικούς ανθρώπους ε, στην Ευρώπη, αν όχι ο κύριος άνθρωπος που ασχολείται με αυτοματοποιημένο ε, αυτοματοποιημένο έλεγχο δεδομένων. Θα σας πει λοιπόν κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο Ανδρέας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας είμαι, αισθάνομαι πολύ αμήχανα όταν γύρω μου κάθονται τόσο διακεκριμένοι ομιλητές. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι στο ύψος. Ε, χαίρομαι που ενδιαφέρεστε για αυτά που έχω να σας πω. Θα ήθελα να σας πω τι κάνουν οι ελεγκτές των δεδομένων. Ας πούμε έχουμε μία δήλωση ότι το ε, Ηνωμένο Βασιλείο έχει 10 φορές περισσότερους μετανάστες από την Ιταλία. Ένας ε, δημοσιογράφος ας πούμε θα πάει σε διάφορους πίνακες ας πούμε και θα κοιτάξει τους αριθμούς των μεταναστών ανά χώρα, ανά κτλ. Και έχει γίνει αυτός ο έλεγχος. Ήταν λάθος αυτός ο χειρισμός, δεν υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Ε, θα έχετε ήδη ακούσει ε, ότι ζητείται όλο και περισσότερο έλεγχος δεδομένων. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε όλο και περισσότερες ιστοσελίδες που κάνουν αυτή τη δουλειά τα τελευταία χρόνια. Το 2010 ε, αναφέρθηκε, το 1710 συγγνώμη αναφέρθηκε ότι τα ψεύδια ας πούμε ε, πάνε πολύ μακριά ε, και η αλήθεια ακολουθεί. Αυτό το 1710. Ε, είναι πολύ εύκολο να διαδοθούν ψευδείς ειδήσει. Πριν, πριν σας μιλήσω πώς γίνεται αυτόματα αυτό το θέμα, είναι, ε, λειτουργεί, θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, έχουν γίνει μελέτες που λένε ότι μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ. Αν πει σε κάποιον ότι αυτό που πιστεύει είναι λάθος, ε, θα πιστεί ακόμα περισσότερο για αυτό που πιστεύει. Ε, λόγω του ότι έχει διαβάσει κάποια πράγματα σε αυτές τις προκατηλημένες ιστοσελίδες. Ε, ή έχουμε δει, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι διαβάζουν διορθώσεις ειδήσεων και όμως δεν αλλάζουν την άποψή τους. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι λειτουργεί, αλλά χρειάζεται και χρόνο και προσπάθεια. Ε, εδώ σας αναφέρω δύο μελέτες, μία στην, για ψυχολογικά θέματα και μία για την πολιτική. Και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε ότι χρειάζεται χρόνος, δεν γίνεται ε, αυτόματα. Ε, χρειάζονται διάφορα αποδεικτικά στοιχεία για να αρχίσει να πιστεύει λιγότερο ο, ο κόσμος κάτι ψευδές. Ας πούμε, Κάποιοι έχουν, πιστεύουν ας πούμε σε UFO ας πούμε. Ε, αυτό δεν τους επηρεάζει την καθημερινότητά τους και χρειάζεται να γίνει πολλή προσπάθεια για να μειωθεί αυτή η πίστη τους σε ψευδείς ειδήσει. Ε, ας πούμε εγώ είμαι μια, ε, ένας ειδικό ε, στην εκμάθηση της μηχανής. Θα έχετε α, ακούσει ότι μπορεί το μηχάνημα ας πούμε, να γνωρίζει γάτες ας πούμε, φωτογραφίες κτλ. ανάλογα με την ένταση των πιξελών. Ε, θα μπορούσαμε μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τη μηχανή για να κάνει τέτοιες αναγνωρίσεις. Είμαστε επιτυχείς ε, σε αυτό το επίπεδο. Ας δούμε τώρα ε, αν μπορούμε να χτίσουμε ένα μηχάνημα το οποίο να κάνει αυτό που κάνουν οι άνθρωποι, ας πούμε. Ε, αυτό, αυτή ήταν η σκέψη. Ε, με τον Σεμπάστιαν από το 2014 αρχίσαμε να σκεφτόμαστε. Τι θέλουμε ας πούμε από, την αυτοματοποιημένη, από το αυτοματοποιημένο έλεγχο των δεδομένων. Καταρχάς θέλουμε ε, διαφάνεια των αλγορίθμων. Θέλουμε... Δεν αρκεί να μας πει ε, το μηχάνημα είναι αλήθεια ή είναι ψέμα. Αυτό που θέλω να δω είναι και μια δικαιολογία και κάτι άλλο που έχει αναφερθεί είναι ότι θα πρέπει να μπορούμε να τσεκάρουμε το κατά πόσο είναι σωστό κάτι άλλο. Δεν αρκεί να πούμε σωστό ή λάθο. Τα μοντέλα του ή άλλω θα κάνουν λάθη. Ε, είναι σημαντικό να μαθαίνουν από τα λάθη του. Ε, για να μην χρησιμοποιούμε ψευδεί πληροφορίε για τι αποφάσει μα. Επίση, ε, η γενίκευση σε διάφορου ε, τομεί. Α πούμε, ε, ανέφερα ήδη τη μετανάστευση. Υπάρχουν και άλλοι τομεί. Ε, η οικονομία, η υγεία, ο αθλητισμός. Ανδρέα, σε παρακαλώ πιο αργά, γιατί έχουμε χρόνο. Λίγο πιο αργά. Πρώτη φορά με μεταφράζουν και γι' αυτό είμαι αγχωμένος. Θα πιω λίγο νεράκι για να χαλαρώσω. Οι φίλοι μου που κάνουν τέτοια δουλειά μου είπαν ότι θα πρέπει να βάλω και ενδιαφέροντα μορφολογικά φαινόμενα στην ομιλία μου. Ε, έχω ένα προβληματάκι με την ταχύτητα, όπως καταλάβατε. Για να δούμε αν η μηχανή θα μπορούσε να σε μεταφράσει. Δύσκολο θα ήταν και με τη μηχανή. Σας έλεγα λοιπόν ότι προσπαθούμε να κάνουμε γενικεύσεις, να περάσουμε σε διάφορους τομείς, οικονομία, υγεία, αθλητισμό. Και το τελευταίο που είναι σημαντικό είναι όταν κάνουμε ε, αναγνώριση εικόνων ή μεταφράσεις, ε, έχουμε επιτυχίες γιατί βασιζόμαστε, για να κάνουμε την κατάρτιση, ας πούμε, την εκπαίδευση της μηχανής, σε πάρα πολλά δεδομένα. Μιλάμε για πολλά δεδομένα και η μετάφραση μίας πρότασης μπορεί να χρειαστεί χρόνο, αλλά δεν χρειάζεται μια ολοκλημέρα, ας πούμε, κατά μεσόρο. Ε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τόσα πολλά δεδομένα ε, όπως αυτά που χρησιμοποιούμε για, για την αναγνώριση εικόνων, ας πούμε, βάσει τις πιξέλες κτλ, για να κινηθούμε τόσο γρήγορα και στον έλεγχο των δεδομένων. Λοιπόν, καταρχά, ακούμε, ας πούμε, ισχυρισμού, ότι ε, οι Σύριοι πρόσφυγες, ας πούμε, μόλις έρθουν ε, στην Αμερική δεν τους ελέγχει το FBI, ας πούμε. Σωστό ή, αλήθεια, ή ψέμα. Αυτή είναι μια γνώμη. Δεν μπορούμε να πούμε αλήθεια ή ψέμα. Τι σημαίνει ότι δεν ελέγχεσαι, α πούμε. Μπορούμε να το συζητήσουμε, α πούμε. Δεν του ελέγχει του πρόσφυγε κανεί. Θα μπορούσε να είναι μια συμφωνία που υπάρχει, α πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε αλήθεια ή ψέμα. Επίσης, ε, υπάρχουν ε, κάποιοι άλλες, κάποιες, ε, κάποιοι κάποιες ε, Δεν μπορούμε να πούμε πάντα σωστό ή λάθος. Αν έβαζα, ας πούμε, φωτογραφίες πολιτικών ή άλλων σημαντικών ανθρώπων, ας πούμε, θα, σας, ε, θα είχε σημασία για σας. Πιστεύω ότι ναι. Γιατί επηρεαζόμαστε όλοι. Αλλά το θέμα αυτό ακριβώς είναι. Ε, το πρόβλημα ακριβώς αυτό είναι. Δεν θα έπρεπε να βάζουμε εκεί φωτογραφίες. Γιατί όλοι μας, και εγώ ακόμα, μπορούμε να παραπλανηθούμε από κάποιον που εμπιστευόμαστε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κόσμο μα λέει ψέματα γιατί θέλει να μα εξαπατήσει ντε και καλά. Συμβαίνει και αυτό, αλλά όχι πάντα. Είναι πολύ σημαντικό να, το να αγνοήσουμε το ποιος το λέει και να εστιάσουμε στο τι λέει ακριβώς. Επίσης, εάν κάποιος χρησιμοποιεί προχωρημένο λεξιλόγιο, ε, σημαίνει ότι αυτά που λέει είναι πιο αληθινά, πιο σωστά. Ούτε αυτό ισχύει, γιατί μπορεί κάποιο να πει αλήθεια μιλώντας πολύ πολύ απλά. Ε, μπορεί να μην είναι τόσο ομορφωμένο, αλλά μπορεί να μην ψεύδεται όμως. Άρα, τι κάναμε λοιπόν μια πρώτη προσπάθεια το 2015. Ε, πήραμε πολύ απλούς ισχυρισμού. Ας πούμε ε, το Λεσόθο που είναι μια, ένας στην, κοντά στην Νότια Αφρική έχει ένα πληθυσμό 2 εκατομμύρια ας πούμε. Ε, α, πάμε λοιπόν σε διάφορα, και ψάχνουμε διάφορα στοιχεία να δούμε ποια είναι η απάντηση. Σπάσαμε το κομμάτι σε δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα προσπαθούμε να δούμε Πού είναι οι δηλωσει σε αυτόν τον ισχυρισμό. Σε αυτή την πρόταση μιλάμε ότι είναι η χώρα το Λεσόθο, ποιο είναι ο πληθυσμό και λέμε ότι ο πληθυσμό είναι 2 εκατομμύρια. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Στο δεύτερο βήμα είναι να πάμε στι βάσει δεδομένων τη Παγκόσμια Τράπεζα, να δούμε τι νούμερο υπάρχει εκεί για τον πληθυσμό και να επαληθεύσουμε το ποσοστό σφάλματο. Πόσο μακριά είμαστε από το νούμερο που υπήρχε στη βάση των δεδομένων. Αυτό ικανοποιεί αυτά που θέλω εγώ από τον αυτοποιημένο έλεγχο. Καταρχά είναι πολύ απλό, αλλά καταρχά υπάρχει διαφάνεια. Σα σας λέω, α πούμε, το λάθο το λάθος είναι 0,09 και όχι 0,5, Φερρυπίν. Δεν θα σα πω καν ότι είναι σωστό ή λάθο εδώ. Σα λέω 0,09. Και εσύ ω χρήστη θα πρέπει να αποφασίσετε αν είναι ένα ε, αποδεκτό επίπεδο ακρίβεια ή όχι αυτό. Σα το αφήνω σε εσά. Δεν θα σας πω καν είναι σωστό ή λάθο. Το τελευταίο είναι ότι μάθαμε χωρίς δεδομένα για κατάρτιση. Κανένας δεν πήγε δηλαδή με διάφορες φράσεις να λέμε ότι ε, αυτός ο ισχυρισμός ή τον πληθυσμό είναι αλήθεια ή ψέμα. Γίνεται αυτόματα. Σας λέω το, έτσι σχηματικά την ιδέα. Υπάρχουν πολλά πράγματα από πίσω. Τι κάναμε λοιπόν. Πήραμε έναν υπολογιστή μια μικρή εφαρμογή, διάβασε πάρα πολλά κείμενα από το ίντερνετ και βρήκε προτάσεις που μιλάνε για χώρες και νούμερα. Έτσι. Για τον πληθυσμό θα μπορούσαν αυτά νούμερα ή για διάφορα άλλα πράγματα, τουρίστες ε, που επισκέπτονται τη χώρα, ας πούμε, οτιδήποτε. Και από εκεί κάναμε ένα πίνακα και σε αυτό το πίνακα, καταρχάς, πάνω-πάνω, έχουμε τις, πληροφορίε πληροφορίες από τις βάσεις ε, δεδομένων, το σωστό, ας πούμε, πληθυσμό για τη Γαλλία, την Ισλανδία και τη Ρωσία. Και έχουμε και κάποια pattern το, το πώς υπάρχουν, ε, ποια λέξη ακολουθεί την άλλη, ας πούμε τι pattern έχουν και βλέπουμε ότι οι ισχυρισμοί είναι πολύ κοντά σε αυτά που λένε οι βάσεις δεδομένων. Έτσι βρίσκουμε κάποια pattern για το πώς ε, εκφραζόμαστε σε διάφορες γλώσσες. Επίσης, το τρίτο είναι ε, ο, τα ποσοστά πληθωρισμού, που είναι συνήθως μικρά νούμερα. Ε, και βλέπεις εδώ πέρα ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Έτσι. Το κομπιούτερ βέβαια δεν, δεν καταλαβαίνει καθόλου τις διάφορες λέξεις, τις διάφορες γλώσσες. Κοιτάει τα νούμερα. Προσπαθούμε να βρούμε λοιπόν ισχυρισμούς που δεν έχουν την ε, λέξη πληθυσμός. Όταν λέει ο πληθυσμό είναι τα τόσο, α πούμε, είναι εύκολο. Αλλά μερικέ φορέ μιλάει για κατοίκου ή για χρησιμοποιεί άλλε λέξει. Ή η διαδοχή των λέξεων, ας πούμε, ε, όταν εμφανίζεται με την ίδια διαδοχή, ας πούμε, με αυτή που υπάρχει στη βάση δεδομένων, είναι πολύ εύκολο για το μηχάνημα. Και βλέποντας τέλος πάντων πολλά δεδομένα, βλέπουμε ότι ε, όταν λέμε ότι η Γαλλία ε, έχει τον ίδιο αριθμό τουριστών με τον πληθυσμό της, ας πούμε, ε, μπορούμε να καταλάβουμε ε, αν είναι σωστό ή λάθος αυτό. Έτσι καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το πράγμα. Μπορείτε να συγκρίνεται pattern, διάφορα μοντέλα ας πούμε. Το θέμα είναι, λειτουργεί αυτό το πράγμα. Κάναμε... Κάναμε διάφορους συσχετισμούς, ε, συλλέξαμε 100.000 ε, σελίδες και βρήκαμε τι ποσοστό ε, ακρίβειας υπάρχει, 60% καλή είναι, αλλά θα μπορούσε να βελτιωθεί. Στο δεύτερο, στη δεύτερη φάση κάνουμε μια επαλήθευση. Είπαμε, εντάξει, εάν ο αριθμό είναι σωστό, α πούμε, έχει, λέει σωστά ποιο είναι ο πληθυσμό και εκτιμά, α πούμε, το λάθο, ε, τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι σωστό ή λάθο αυτό που λέει. Γιατί δεν έχουμε βάση δεδομένων με στοιχεία σωστό ή λάθο. Στην πραγμότητα, ε, αυτό που βρήκαμε βρήκαμε ότι ο κόσμος χρησιμοποιεί πεπαλαιωμένα στατιστικά δεδομένα. Χρησιμοποιούνται συχνά ξεπερασμένα στατιστικά στοιχεία για να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις. Αλλά γίνονται και λάθη. Το άλλο που κάναμε είναι να κοιτάξουμε διάφορες πηγές που υποστηρίζουν ε, ή καταρρύπτουν κάτι. Ε, Παραδείγματο χάρη, εδώ πέρα λέμε ότι οι γιατροί επιβεβαιώνουν την πρώτη περίπτωση θανάτου από γενετικά τροποποιημένη ε, τροφή. Ε, ε, οι δημοσιογράφοι βρήκαν ότι είναι λάθος αυτός ο ισχυρισμός. Ε, η μία πηγή που είναι κατά της του ισχυρισμού, δηλαδή που καταρρύπτει τον ήθο, την επισκέφτηκαν μόνο 15, 1.500 περίπου άτομα. Ενώ τον αθασμένο ισχυρισμό τον επισκέφτηκαν 60.000 άτομα. Και παρότι ας πούμε, οι δημοσιογράφοι κάνουν ό,τι μπορούν για να διορθώσουν τα πράγματα, η ζημιά έχει γίνει γιατί ε, χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο τα ψευδή στοιχεία ε, παρά ε, η κατάρριψη του ισχυρισμού, ας πούμε. Δηλαδή ο κόσμος δεν πάει να επισκεφθεί την, ε, τις ιστοσελίδες που καταρρύπτουν τον ισχυρισμό. Επίσης, κάναμε μία αυτοματοποιημένη κατά, κατάταξη της, ε, της τάσης των ανθρώπων και βρήκαμε ότι υπάρχει ακρίβεια 73%. Επίσης, ε, ασχοληθήκαμε και με, τα, με τις ψευδείς ειδήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Να υπάρξουν, να βρεθούν, ε, να συσταθούν καλές ομάδες για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Υπάρχουν 300 ισχυρισμοί από ιστοσελίδες που καταρρύπτουν ε, ψευδείς ειδήσει. Μαζί με τους αδέλφους από το Amazon Research προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία βάση δεδομένων με πάρα πολλούς ισχυρισμούς, 100.000 ισχυρισμούς και να φτιάξουμε ένα αλγόριθμο που να λέει αυτό, γι' αυτό υπάρχουν ε, στοιχεία. Ε, το θέμα είναι όμως να παραπέμπουμε και στις πηγές. Πού το βρήκαμε αυτό στην Wikipedia κτλ. Και, και αυτό θα το δημοσιεύσουμε. Μετά την έρευνα, τι θέλουμε να κάνουμε. Ή να φτιάξουμε ένα, μια ιστοσελίδα όπου οι χρήστες θα μπορούν να τσεκάρουν αυτόματα οτιδήποτε θέλουν, οποιονδήποτε ισχυρισμό. Ε, ελπίζουμε και οι χρήστες να μας δίνουν και κάποια, να μας τροφοδοτούν, ας πούμε, κάποιες απόψεις. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να μάθουμε και να βελτιώσουμε και τα μοντέλα μας. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα σε εμά και σε αυτούς που κάνουν έλεγχο τους ανθρώπους, δηλαδή τους ελεγκτές που το κάνουν χειρονακτικά. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια διαφορετική σχέση ε, και να δώσουμε ένα προϊόν που θα είναι χρήσιμο στην εποχή των, ε, της χιονικής δικτύωσης. Ε, ούτω ώστε να μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία στο ίντερνετ, ούτω ώστε ο κόσμος να πρέπει να σκέφτεται δύο φορές αν θα θα πει κάτι ψευδές. Επίσης, δεν θέλω να φτιάξω έναν αλγόριθμο που θα μου λέει αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Θέλω να εκπαιδεύσω το κοινό από πολύ νεαρή ηλικία, από τα παιδιά του δημοτικού, για να τσεκάρουν τα παιδιά από μόνα τους και να αποφασίζουν από μόνα τους αν είναι κάποιος ισμόστό ή σωστό ή λάθο. Ε, αναφέρθηκε πολύ η υγεία, οι πληροφορίε για την υγεία είναι πολύ σημαντικές. Γιατί σήμερα, αντίθετα από 10-20 χρόνια πριν, το πρώτο πράγμα που, αισθάνομαι, που κάνω όταν είμαι άρρωστο ή αισθάνομαι άρρωστο δεν είναι να πάω στο γιατρό, αλλά να ψάχνω στο Google. Και ε, ψάχνω να βρω πληροφορίε. Υπάρχουν πληροφορίε, υπάρχουν πληροφορίε, μόνο που πρέπει να τι ελέγξει κανεί. Ευχαριστώ. Thank you, uh, uh, Είσαστε ζωντανή, ε, ζωντανό παράδειγμα ότι ότι χρειάζονται ακόμα ε, διερμηνείς, φυσική παρουσία διερμηνέων. Σχετικά τώρα με τα δεδομένα που έχουν σχέση με ιατρική. Οι αλγόριθμοι μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη παρέμβαση και αυτό είναι επικίνδυνο ή όχι. Όσον αφορά τις κατασκευασμένες ειδήσει στον αγώνα μεταξύ ανθρώπων και μηχανών, τελικά οι άνθρωποι κερδίζουν. Το ερώτημά σας είναι κατά πόσον οι άνθρωποι μπορούν να νικήσουν τις μηχανές. Εξαρτάται ε, εάν πρόκειται για σκάκι, ενδεχομένως ε, να μπορούν να νικήσουν, αλλά όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, Κατ' ουσία μπορούμε να βρούμε παραδείγματα όπου καταδεικνύουν ότι δεν μπορεί να παραπλανηθεί κανένας άνθρωπος. Βέβαια, έχουν υπάρξουν έρευνες για τον εντοπισμό παραπλάνησης και βλέπουμε ότι ο ανθρώπινος νους και η ανθρώπινη παρέμβαση είναι πολύ πιο αξιόλογοι από τον αλγόριθμο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μία συνεργασία, η μία πλευρά αλληλοσυμπληρώνει την άλλη. Πολύ ωραία. Ο κύριος Τζον Στίνμπερκ από τη Google θα λάβει τώρα το λόγο. Είναι manager για public policy στην Ευρώπη. Ήρθε από τις Ηνωμένε Πολιτείε και έχει εργαστεί σε διάφορες πολιτικές εκστρατείες στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ξέρω ότι έχετε χάσει βέβαια μία. Φαντάζομαι ότι ε, γνωρίζετε καλά τον κλάδο σα. Εγώ εργάζομαι κυρίως ε, σε πολιτικές εκστρατείες, πράγματι έχω χάσει μερικές. Είναι μεγάλη χαρά για μένα το ότι μπόρεσα να έρθω σήμερα εδώ, να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Οι συζητήσεις που είχαμε μέχρι τώρα ε, πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακέ και ε, πολλές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που βασίζονται σε τεχνογνωσία, σε δεδομένα, σε γεγονότα προσβλέπω στην όλη αυτή τη συζήτηση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι στην Google εμείς σκεφτήκαμε το πώς μπορεί κανείς ε, να αξιολογήσει τις πληροφορίες, τις κατασκευασμένες ειδήσει. Αυτό είναι ο στόχος μας, γιατί και αυτό θα καθορίσει πώς εμείς οι μηχανικοί θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Ο στόχος μας λοιπόν είναι οι πληροφορίες να είναι γενικώ προσπελάσιμες. Και όπως αλλάζει το διαδίκτυο, όχι κάθε χρόνο, αλλά κάθε μέρα, ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος. Το θέμα είναι, εξελίσσεται βέβαια και ο στόχος μας. Λίγο χρόνο έχω, τρία πράγματα θα δείξω. Ε, πρώτον, πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα, πώς οι αλγόριθμοι οργανώνουν την πληροφορία, πως ε, τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση των κατασκευασμένων ειδήσεων και μετά θα αναφέρω και ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να προτρέχουμε στη σκέψη μας και πώς ε, οι άνθρωποι ε, κατακλείζονται κυρίως με πληροφορίες και τελικά πώς λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις. Όσον αφορά καταρχήν την αναζήτηση. Υπάρχουν, θα έλεγα, εκατομμύρια σελίδων με πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Άρα πώς θα βρούμε ποια πληροφορία μας ενδιαφέρει. Όλα αυτά ξεκινάνε ε, και πριν ξεκινήσουμε, δηλαδή με το να ψάχνουμε σε διάφορους ε, καταλόγους. Έχουμε συγκεκριμένες μηχανές ε, οι οποίες οργανώνουν όλα αυτά και όταν καταλήξει κανείς σε κάποια ιστοσελίδα τότε ε, βλέπουμε ότι εντοπίζονται κάποιες λέξεις κλειδί. Εμείς αυτά τα ταξινομούμε τι γίνεται όταν κάνει κανείς μία αναζήτηση. Μιλάμε για εκατομμύρια ιστοσελίδες και πάρα πολλές απαντήσεις. Το δικό μας το σύστημα της ταξινόμησης ψάχνει όλες αυτές τις σελίδες για να σας δώσει τα σωστά και χρήσιμα αποτελέσματα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτά τα συστήματα της ταξινόμησης βασίζονται σε μία σειρά αλγορίθμων οι οποίοι αναλύουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Και στις συζητήσεις που έχουμε σχετικά με την αναζήτηση, νομίζω είναι σημαντικό να έχει κανείς κατά νου ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο χρήστης. Εμάς μας ενδιαφέρει να προσφέρουμε σημαντικές πληροφορίες και μας ενδιαφέρει επίσης να βελτιώσουμε τις δυνατότητες που έχουμε στο να σας προσφέρουμε χρήσιμες πληροφορίες. Κάνουμε λοιπόν αλλαγές συνεχώς, ε, διότι εμεί πιστεύουμε ότι η αναζήτηση δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ως πρόβλημα. Και πραγματικά θα σε εκπλήξει πώς οι μηχανικοί καθημερινά ασχολούνται με την αναζήτηση. Μόνο το 2006 είχαμε 150.000 περίπου πειράματα για αλλαγές στην αναζήτηση ε, Αυτά μόνο το 2016, διότι οι μηχανικοί μας έχουν πάρα πολλές ιδέες ε, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, προσφορά μας. Βασιζόμαστε επίσης σε πάρα πολλά τεστ που αφορούν στον καταναλωτή. Προσπαθούμε να αναλύσουμε τις μήτρες ε, και πώς θα προτείνουμε συγκεκριμένες αλλαγές. Έχουμε ε, και αναγνώστες ε, που εξετάζουν ε, διάφορα αποτελέσματα, προσπαθούν να δούνε πώς μπορεί να αναζητηθεί η καλύτερη πληροφορία. Κάνουμε επίσης και Taste Live, όπου Αυτά λέγονται test ABC, δηλαδή χρησιμοποιούμε τους χρήστες σε σχέση με το αποτέλεσμα. Προσπαθούμε να δούμε ποιο αποτέλεσμα παίρνει περισσότερα κλικ και τέλος εξυπηρετούμε και τους χρήστες μας με την έννοια τους ε, ρωτάμε και για νέα χαρακτηριστικά. Κάθε φορά λοιπόν όλα αυτά μπαίνουν στις ε, μηχανές και όπως σας είπα έγιναν 150.000 πειράματα. Ε, κάναμε πάρα πολλούς πειραματισμούς Αν θέλετε μπορώ να μπω και σε περισσότερες λεπτομέρειες δύο λεπτά, αλλά θα, σας, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω πώς προσπαθούμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση των κατασκευασμένων ειδήσεων. Αυτό για μας είναι μια γνωστή πρόκληση. Είναι μια μορφή spam. Ε, είναι προσπάθεια να χρησιμοποιούμε αλγορίθμους για να αντιμετωπίζουν το χαμηλό, χαμηλής ποιότητας αποτέλεσμα. Εμείς πριν από 20 ε, περίπου χρόνια ως Google αρχίσαμε να ασχολούμαστε με αυτό και το εξακολουθούμε και σήμερα. Γιατί τα αποτελέσματα της αναζήτησης δεν είναι χρήσιμα αν δεν μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε. Ε, θα μιλήσω λοιπόν για τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να βρουν ποιοτικό περιεχόμενο. Και έχει νόημα να υπενθυμίζουμε στους ανθρώπους γιατί η Google ε, είναι στην πρώτη θέση στη μηχανή αναζήτησης. Ε, εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι οι άνθρωποι αναζητούν πληροφορίες, άρχισαν να ζητούν πληροφορίες για το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου ε, στη, με βάση την επίθεση της 11 ε, Σεπτεμβρίου. Ε, ποιος ήταν ε, ο αρχιτέκτονας, πότε κατασκευάστηκε το κτίριο. εκείνη όμως την ημέρα οι άνθρωποι δεν τους ενδιαφέρε αυτό ακριβώς. Έτσι λοιπόν οι μηχανικοί μας θέλησαν να δώσουν μια καλύτερη νήση και έτσι πρόκειται το Google News. Ε, συγκεντρώνουμε πληροφορίες από πάρα πολλές πηγές ανά τον κόσμο, ε, τα εντάσσουμε στα Google News ε, ε, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία προσαρμόζονται έτσι ώστε να υπάρχει μια ποιοτική έρευνα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αποκρύπτονται πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες, με τους στόχους, ε, να υπάρχει ανάλυση πρόσφατων γεγονότων, να υπάρχει λογοδοσία, βιογραφικά και επίσης θα πρέπει να περιορίζεται και ο αριθμός των παραπλανητικών παρεμβάσεων. Εμείς δεν απορρίπτουμε πηγές λόγω ιδεολογικών απόψεων. Ε, ο στόχος της Google News είναι να οδηγεί τους καταναλωτές σε συγκεκριμένα websites ε, όπου εκεί μπορούν και οι ίδιοι να ελέγχουν το περιεχόμενο. Δέκα δις ε, το μήνα σε συγκεκριμένους εκδότες στις ιστοσελίδες τους δωρεάν και μετά αυτό αξιολογείται ε, αξιολογείται και κοστίζει αυτό το κλικ. Ε, επίσης ε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους εκδότες να εκμεταλλεύονται οικονομικά αυτά τα κλικ. Έχουμε και μια νέα δυνατότητα, προσφέρουμε μεγαλύτερη ευηλιξία στους εκδότες για να πείθουν καλύτερα τους χρήστες να καταφεύγουν στις δικές τους τις εκδόσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια είναι όπως σας είπα ποιοτικό περιεχόμενο και γι' αυτό το λόγο έχουμε πριν από λίγα λόγια εισαγάγει την πρωτοβολία Google News. Ε, μέχρι τώρα έχουμε προσφέρει ε, χρηματοδότηση για πάρα πολλά προγράμματα με βάση τα έσοδά μας. Ε, προσφέρουμε χρήματα όχι μόνο στους εκδότες αλλά Έχουμε συνεργασία και άμεση συνεργασία με τους εκδότες, κυρίως για χρήστες που αναζητούν πληροφορίες στα κινητά τους τηλέφωνα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους εκδότες, όπως σας είπα, να κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Επίσης, ε, συνεργαζόμαστε όχι μόνο επιχειρηματικά. Έχουμε μία ομάδα η οποία μας βοηθάει ε, σχετικά με τον έλεγχο των δεδομένων και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι προσφέρουμε και δωρεάν πρωτοβουλίες. Στηρίζουμε οργανώσεις ε, ε, οι οποίες έχουν προκύψει για να υπάρχει η βέλτιστη πρακτική. Και έτσι καταλήξαμε σε συγκεκριμένες ε, αναλύσεις για εκλογές που έγιναν στη Γαλλία, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και εξετάζουμε και διάφορα προγράμματα με ε, μη κυβερνητικού οργανισμούς. Ο στόχος μας είναι να αναζητήσουμε λύσεις ε, για ποιοτική ε, δημοσιογραφία. Πρόσφατα λοιπόν δημοσιεύτηκαν ε, κάποιες ε, συγκεκριμένες αρχές. Αυτό έγινε συγκεκριμένα την ε, προηγούμενη εβδομάδα. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος των γεγονότων είναι απολύτως απαραίτητος για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την πρόκληση των κατασκευασμένων ειδήσεων. Πρόσφατα με μια άλλη εταιρεία δώσαμε τη δυνατότητα στους εκδότες στα Google News να έχουν μια ειδική ετικέτα που επιστρέφει επιτρέπει τον έλεγχο των γεγονότων και έτσι οι αναγνώστες μπορούν να ελέγχουν τα γεγονότα. Στις αρχές αυτού του έτους ανακοινώσαμε ότι αυτές τις ετικέτες θα τις επεκτείνουμε και στις, σε άλλους τομείς, όχι μόνο στα Google News, ε, αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι ε, συνεργαζόμαστε με εκδότες και με οργανώσεις ε, που κάνουν τον έλεγχο. Εμείς τους προσφέρουμε τα απαραίτητα εργαλεία. Διεπιστώνουμε επίσης ότι όλα αυτά αλληλοσυμπληρώνονται. Για μας αυτό που έχει σημασία είναι ο ρόλος που μπορεί να τριματίσει η Google. Πρόσφατα έγινε και μία μελέτη που κατέδειξε ότι οι ερευνητές χρησιμοποιούν τον έλεγχο των γεγονότων, άρα δηλαδή διαβάζουν κάτι στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, τα ακούνε από φίλου ή από πολιτικού τηλεόραση και μετά ελέγχουν κατά πόσο αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει υπάρχει έλεγχος των γεγονότων. Επίσης πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση ακολούθησε το χρήμα και αυτό βοηθάει ε, να αντιμετωπιστούν οι κατασκευασμένες ειδήσει. Γιατί αν δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο ε, τότε δεν υπάρχει και λόγος ε, για τις ε, κατασκευασμένες ειδήσει. Γι' αυτό το λόγο εμείς ε, αποφασίσαμε ότι αν κάποιοι εκδότες ε, προσφέρουν fake news, αυτοί θα αποκλείονται από τη συνεργασία μας. Δηλαδή θέλουμε να μην προσφέρουμε κοινωνικά κίνητρα και το 2016 εμείς αφαιρέσαμε 1,7 δισεκατομμύρια καταχωρήσεις ε, γιατί παραβιάστηκε η πολιτική μας. 100.000 ε, εκδότες ε, διαγράφηκαν και περίπου 3 εκατομμύρια βίντεο τα απαγορεύσαμε και αυτά. Όπως σας είπα, εμείς στραφήκαμε κατά πολλών ιστοσελίδων με κατασκευασμένες ειδήσει. Ε, πολλές φορές για ποιοτικού λόγους επιλέγουμε να μην ε, επιλέξουμε μία καταχώρηση. Και ε, αναφέρομαι και σε ομιλίες κηρύγματα μίσους, ε, ε, σε πάρα πολλά παρεμφερή αλλά και σε σελίδες ας πούμε, που προάγουν το hacking. Αυτό που ενδιαφέρει ο τέταρτος τομέας είναι το τι κάναμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να αναλάβουμε δράση. Κάναμε κάποιες αλλαγές τον Απρίλιο. Το πρώτο είναι ότι έχουμε ένα feedback. Αναγνωρίσαμε, αναγνωρίζουμε ότι ορισμένα από τα προϊόντα μας ε, ε, δεν εκπλήσουν. Μερικές φορές ε, ε, οδηγούν σε απρόσμενα αποτελέσματα. Ε, Παραδείγματο χάρη είναι ε, όταν μπαίνει κανείς στη Google, ίσως μπορεί κανείς να προβλέψει τι ακριβώς θα δει. Ε, ως εκ τούτου βλέπουμε ότι πολλές φορές μπορεί κανείς ε, να αποφύγει ορισμένες προκλήσεις. Επίσης, μπορεί κανείς ε, να ε, έρθει σε επαφή με εμά, να μας ενημερώσει σε σχέση με το περιεχόμενο. Αυτό το feedback το χρησιμοποιούμε για να έχουμε καλύτερους αλγόριθμους και επίσης ε, θέλουμε και να αλλάξουμε την αξιολόγηση των αλγορίθων μας. Αυτό σε σχέση με τα αποτελέσματα. Και ένας τρόπος που το κάναμε αυτό για να ε, εκπαιδεύσουμε καλύτερα τους αλγορίθμους εισαγωγικά είναι να εκδώσουμε οδηγίες ε, που υπάρχουν, όπως σας είπα, και εξηγούν τα αποτελέσματα. Δεν είναι απλά απορίσματα, αλλά πρόκειται για συγκεκριμένα αποτελέσματα που προβάλλουμε για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε ε, περιεχόμενο υψηλού επίπεδου. Και αυτό νομίζω ότι βοηθάει τους μηχανικούς μας να αξιολογήσουν καλύτερα τους αλγορίθμους και το τι διαδραματίζεται κάθε μέρα. Αυτό επίσης ε, που θέλω να σα πω είναι ότι σχετικά με τι οδηγίε, ξέρουμε ότι οι οδηγίε αυτέ δεν ήταν αποτελεσματικέ στο να αξιολογήσουν λάθο ε, ειδήσει. Εμάς μας ενδιαφέρει ε, το αποτέλεσμα να είναι ακριβές, υψηλή ποιότητα, γιατί αν δεν εξυπηρετήσουμε τέτοιου είδους στόχους, ε, ε, κατ' ουσίαν και εμεί θα προβάλλουμε κατασκευασμένε ειδήσει και καταλαβαίνετε ότι αυτός δεν είναι ο στόχος μας, γιατί πρόκειται για στελίδες ε, που είναι ε, καταξιωμένες. Για μας αυτός είναι ο στόχος μας. Έχουμε το feedback. Το feedback που το χρησιμοποιούμε για τους αλγορίθμους μας έτσι ώστε να έχουμε τις αξιόλογες και σωστές πληροφορίες. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω και το εξή. Ένα εργαλείο το οποίο εισαγάγαμε πρόσφατα και που κατά την άποψή μας ε, βοηθάει να αντιμετωπίσουμε τις τις ε, προκλήσεις ε, δίδοντας ε, σωστές πληροφορίες. Είναι το Google Search App το οποίο παρουσιάσαμε το καλοκαίρι σας. Το έχετε ήδη στο κινητό σας τηλέφωνο. Αυτό είναι. Το βλέπετε. Το Google Search App κάνει το εξής. Ε, αποκαλείται The Feed. Έχετε ένα παράδειγμα εδώ και οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Είτε είναι ειδήσει, αθλητικές ειδήσει, μετοχές, οτιδήποτε. Επιλέγουν λοιπόν το τι τους ενδιαφέρει. Αυτό ε, ενημερώνεται αυτή η ιστοσελίδα, ενημερώνεται από τα δικά τους τα θέματα που τους ενδιαφέρουν τους ίδιους. Και νομίζω ότι αυτό ε, βοηθάει στο να αντιμετωπιστούν τα filter bubbles. Ε, επίσης προσφέρουμε σκόπιμα πολλές πηγές όταν δίδουμε ειδήσει για θέματα που ενδιαφέρουν τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι παίρνουν πληροφορίες από πάρα πολλές πηγές. Οριζόντια αυτή η διαδικασία βλέπετε ότι οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για κάποια είδηση από διάφορα πρίσματα και κάνουμε και έλεγχο των γεγονότων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με μεγάλη χαρά να συμμετάσχω στη συζήτηση. Thanks, John. Um... John. Πολύ ενδιαφέρον να, ακούμε τι κάνει ακριβώς η Google για να αντιμετωπίσει διάφορα πράγματα. Οι δημιουργοί σας δημιουργούν ε, πάρα πολλές ε, έξυπνες μηχανές συλλογή δεδομένων ε, που στοχεύουν εμπορικά μηνύματα. Έτσι βγάζετε λεφτά. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι γιατί αυτοί οι φανταστικοί άνθρωποι δεν σκέφτηκαν από την αρχή ότι η συλλογή δεδομένων μπορεί να έχει και μια σκοτεινή πλευρά και να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένου σκοπού. Γιατί λοιπόν κάποια πράγματα που βάλετε από την αρχή στους αλγορίθμου σα τα βάλατε, α πούμε, ενώ είναι προβληματικά. Πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειε, σε συγκεκριμένα πράγματα. Ε, εάν μιλάμε με γενικολογίε, τελικά δεν, δεν μιλάμε για το πώς λειτουργεί το σύστημα και τι κάνει ο μηχανικός για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα πράγματα. Φερρυπίν, ας πάρουμε ένα τομέα όπου αναγνωρίζουμε ότι δεν τα πάμε καλά. Ε, θέματα ιστορικής φύσεως, ας πούμε. Παραδείγματο χάρη για την, την άρνηση του ολοκαυτώματος. Αυτό είναι άποψη. Έτσι, δεν θα τον υπερασπιστώ σε καμία περίπτωση. Ένα από τα πράγματα που βρήκαμε είναι ότι Λόγω των σημάτων που χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε για το αν ε, μία ιστοσελίδα είναι χρήσιμη ή όχι, είναι το PageRank ε, που χρησιμοποιεί το Google. Δηλαδή διάφορε ιστοσελίδε που συνδέονται μεταξύ του και αυτό μπορεί να είναι ε, σήμα ότι μπορεί να είναι χρήσιμη αυτή η ιστοσελίδα για το ερώτημα που ενδιαφέρει κάποιον χρήστη. Το πρόβλημα, ή ένα από τα προβλήματα σε σχέση με την άρση του είναι ότι υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων που αρνείται το ολοκαύτωμα την ύπαρξή του και θέλει οπωσδήποτε να δημιουργήσει με λύσα ιστοσελίδε που, δημιουργ... που συνδέονται μεταξύ του ε, για να προωθήσουν αυτό το απέσιο περιεχόμενο. Ε, και αυτό εξαπάτησε το σύστημά μα. Δεν είναι ότι εμεί πραγματικά δεν το σκεφτήκαμε. Δεν σκεφτήκαμε κάθε πιθανή ε, αρνητική συνέπεια. Κάθε μέρα προσπαθούμε να προβλέψουμε κάτι τέτοιο. Αλλά μερικέ φορέ το παραδεχόμαστε ότι την πατάμε. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα όπου αλλάζουμε τον αλγοριθμό μας για να προσπαθήσουμε να ε, αξιολογήσουμε καλύτερα και να κατατάξουμε πιο ψηλά ας πούμε, αξιόπιστες πηγές, ας πούμε, μουσεία, Ινστιτούτα κτλ. ή καθηγητές, ούτως ώστε Εάν ψάχνει, α πούμε, γενικέ πληροφορίε για το ολοκαύτωμα, να είμαστε σίγουροι ότι σου δίνουμε χρήσιμε και σωστέ πληροφορίε. Ωραία. Πολύ ωραία. Ο τελευταίο ομιλητή, ο Ρίτσαρντ Άλαν, από το Facebook, που κοιτά την δημόσια πολιτική στην, για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Εγώ τον ξέρω τον Ρίτσαρντ επαγγελματικά εδώ και 25 χρόνια. Δεν σας φαίνεται τόσο γέρος γι' αυτό, αλλά ο Ρίτσαρντ ε, δούλευε ε, στον τομέα της πληροφορικής, ε, επεξεργασία κειμένου κτλ. Είναι παλιός δηλαδή ο Ρίτσαρντ. Σε ευχαριστώ για την εισαγωγή. David, ευχαριστώ τη ΣΤΟΑ για την πρόσκληση και σας εύχομαι καλή τύχη στην αποστολή σας. Θέλετε δηλαδή να ξαναγίνει μοντέρνα η ιδέα το... της κοινωνίας της πληροφορικής. Θα ήθελα εγώ στον χρόνο που έχω να σας μιλήσω ότι υπάρχουν διαφορετικοί αλγόριθμοι. Σε κάθε συσκευή έχει αλγόριθμους ε, στις ε, και συσκευές, ε, στα οχήματα κτλ. Αν το σκεφτούμε πώς πρέπει να αντιδρούν οι θύνοντες, καλό θα ήταν να τους διαχωρίσουμε τους αλγορίθμους. Και οι αλγόριθμοι οι οποίοι μοιάζουν να είναι συγκρίσιμοι, στην πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί. Θα ήθελα να σας δώσω δύο παραδείγματα. Καταρχάς, από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Καταρχάς, ε, κάτι που είναι γνωστό. Δεν θα μιλήσω για τεχνολογία αντισπάμ. Εγώ θυμάμαι, επειδή είμαι παλιός, όταν μπήκε αυτή η τεχνολογία, ακούγαμε διάφορε ιστορίε φρίκης, ότι αυτοί οι αλγόριθμοι θα, από μόνοι τους, ας πούμε, θα, βγάζουν, θα διαγράφουν σημαντικά email. Ενώ σήμερα όλοι ή τέλο 70 ή 80% των email που σας στέλνουν μπαίνει σε, μια, σε ένα κουβά, σε μια ανακαλάθη. Και δεν έχετε κανένα πρόβλημα με αυτό. Και ε, εάν, ας πούμε, ο αλγόριθμος δεν υπήρχε για να σας κάνει την ε, κατάταξη αυτή, δεν θα το ακυρώνατε εσείς αυτό. Θα κάνετε ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, η χρήση των αλγορίθμων για μας είναι, ε, γίνεται ως εξής. Προσπαθούμε να σταματήσουμε τις κακές συμπεριφορές. Και υπάρχει πόλεμος αλγορίθμων ε, μεταξύ, μεταξύ εταιριών όπως εμείς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν τέρατα αλγοριθμικά, ας πούμε, και εμείς προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Η δυσκολία είναι όταν, όταν οι άνθρωποι οι ίδιοι, ας πούμε, κάνουν αυτή τη δουλειά ε, με τον ανυπόμονο ανθρώπινο τρόπο είναι πολύ πιο δύσκολο να το φρενάρουμε αυτό από να διορθώσουμε ας πούμε, τους αλγορίθμους που λειτουργούν σαν αλγόριθμοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, βρίσκονται σε, κάποια, σε κάποιους χώρους, πληρώνονται για να διασπείρουν ψευδείς ειδήσει και εμείς προσπαθούμε να το σταματήσουμε αυτό. Έτσι. Παραδείγματο χάρη, σε όλε τι μεγάλε εταιρείε σήμερα χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι για να ε, σταματήσουν ε, την εμφάνιση πορνογραφικών εικόνων ε, με παιδιά μέσα. Έχουμε μια θαυμάσια τεχνολογία, πολύ καλή, για να σταματήσουμε την παιδική πορνογραφία. Τώρα υπάρχει ενδιαφέρον και από τις κυβερνήσεις ε, και εταιρείε ε, και, συγγνώμη, και φορείς που καταπολεμούν την τρομοκρατία ενδιαφέρονται για αυτά. Ε, υπάρχει ευρεία συνένεση ότι υπάρχει ένα βίντεο προπαγανδιστικό από μια τρομοκρατική οργάνωση με φρικτούς αρκωτηριασμού, ας πούμε. Αν το ε, σταματήσουμε από την, το να διαδοθεί αλγοριθμικά, ε, αυτό γίνεται πολύ πιο γρήγορα από το να πρέπει ο άνθρωπο να σα πει: Κοιτάξτε, τι υπάρχει βίντεο, βγάλτε το, κατεβάστε το, α πούμε. Πάντα όταν το κάνουμε αλγοριθμικά είναι πολύ πιο γρήγορο και καλό. Ε, το πρόβλημα είναι όμω, ακόμα το αναγνωρίζει και στην ανακοίνωσή τη Κομισιόν, είναι ότι υπάρχει τεράστια όρεξη για περισσότερα δεδομένα, όχι λιγότερα δεδομένα. ε, τύπου Snowden, α πούμε. Πολλέ κυβερνήσει λένε θέλουμε κι άλλα, δώστε μα κι άλλα από αυτό το είδο, α πούμε. Και φυσικά εμεί θέλουμε βεβαίω και να προστατεύσουμε την ιδιωτική σφαίρα των ανθρώπων. Ε, Ορισμένε κυβερνήσει μα πιέζουν επίση να μα πούνε. Εάν έχετε, α πούμε, δεδομένα για άτομα τα οποία ανταλλάσσουν τρομοκρατικό περιεχόμενο, δώστε μα τα σα παρακαλώ. Έτσι. Και αυτό είναι θέμα για δημόσια συζήτηση. Αν εμεί βελτιώσουμε λοιπόν του αλγορίθμου για να εντοπίσουμε αυτά τα πράγματα, Πώς αυτό επηρεάζει την σχέση μας με τις διοκτικές αρχές. Αυτή τη στιγμή έχουμε εντοπίσει αυτά τα μηνύματα, ας πούμε. Ε, το κλασικό ας πούμε, στο ίντερνετ είναι ότι η άγνοια είναι ευτυχία. Ας πούμε. Αν δεν, έχεις, δεν ξέρεις κάτι, ας πούμε, έχεις ε, μια κάποιο βαθμό, ένα κάποιο βαθμό αυτόματης προστασίας. Από τη στιγμή που το ξέρεις αρχίζουν να μπαίνουν πολλά ερωτήματα. Υπάρχουν όμως ε, κάποιοι τομείς οι οποίοι δεν δημιουργούν ε, ερωτηματικά και πολεμικές ας πούμε. Έτσι, αυτοί οι τομείς που σας ανέφερα ας πούμε παραδείγματο χάρη, τρομοκρατικό περιεχόμενο, ε, βίντεο του ISIS κτλ. Θέλουμε να τα σταματήσουμε. Επίσης, όταν μας λένε κατεβάστε τα βίντεο του ISIS, φυσικά θα υπάρξουν κάποια ψευδιθετικά. Ε, και η κοινωνία θα πει «Ε, εντάξει, κοιτάξτε, είναι το τιμα που πληρώνουμε, το δεχόμαστε κτλ. Ή η κοινωνία θα κλείσει, α πούμε, θα κατεβάσει ρολά και θα πει δεν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία μέχρι να γίνει τέλεια. Υπάρχει, άλλο Υπάρχει και αυτό το θέμα. Επίση, το πώ θα οργανώσουμε την ε, πληροφορία. Ε, τροφοδοσία με ειδήσει, α πούμε, newsfeed. Ε, Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε εμά και στην έρευνα για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι και πώ κάποιε από τι λύσει που ψάχνει ο, ο, καθένας μπορεί να ποικίλουν. Ε, το καλύτερο σενάριο είναι ένα βιβλιοπωλείο που λέει α πούμε μπαίνω στο βιβλιοπωλείο εγώ και σα δείχνω όλα τα βιβλία για το ποδόσφαιρο. Α πούμε ε, η Google έχει ό,τι βιβλίο έχει γραφτεί από καταβολή κόσμου για το ε, ποδόσφαιρο. Και στην πραγματικότητα σας κάνει ε, όμως. Ένας αλγόριθμος σας προτείνει ε, μία λίστα βιβλίων που νομίζει ότι σας ενδιαφέρουν. Ε, και ε, πρόκειται για βιβλία από ανθρώπων που κάπως είσαστε συνδεδεμένοι, που κάπως σας ενδιαφέρουν. Δεν έχει δηλαδή όλη την πληθώρα ατελείωτων βιβλίων που υπάρχουν. Μόνο των ανθρώπων με του οποίου έχετε κάποια σχέση. Αυτό που βρήκαμε το χρόνο είναι ακόμα και αυτό το περιορισμένο, ο περιορισμένο αριθμό βιβλίων, αν ε, αυξάνεται με το χρόνο. Γιατί συχνά αυξάνουν οι φίλοι σου στο ε, Facebook κτλ. 200-300 κτλ. Και τελικά θα εμφανίζονται πάρα πολλά βιβλία για να μπορέσει να τα διατρέξει όλα. Ε, Επομένω, ο δικό μα ο αλγόριθμο, αυτά τα χιλιάδε βιβλία από του ανθρώπου με του οποίου συνδέεται, ε, στο, τα παρουσιάζει με μια σειρά που θεωρεί ο αλγόριθμο ότι εσένα σε ενδιαφέρει. Πρώτα τα πιο ενδιαφέροντα δηλαδή. Τώρα οι κριτικέ που ακούγονται και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι όχι τόσο η, ο αλγόριθμος ο, ο οποίος παραγγέλει αυτά τα βιβλία, αλλά οι επιλογές που έχεις κάνει στην αρχή. Ορισμένοι επιλέγουν, ας πούμε, κάποια πράγματα. Αν εγώ, ας πούμε, ενδιαφέρομαι μόνο για την Guardian, δεν πρόκειται να ακούσω ποτέ ειδήσει από την Daily Mail, ας πούμε. Θα τις ακούσω ίσως από φίλους, αλλά όχι από το Facebook. Ε, εμείς θα πρέπει να αλλάξουμε τις επιλογές για αυτούς τους ανθρώπους, θα πρέπει να τους προσφέρουμε μεγαλύτερη επιλογή ε, οι προλαλήσαντες ακριβώς έκαναν τέτοια σχόλια προς αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ δεν θέλω να τα κρίνω αυτά. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Αν πούμε σε μια εταιρεία, α πούμε. Κοιτάξτε, στο Facebook υπάρχουν ανησυχίε για μα ότι είμαστε πάρα πολύ ισχυροί και από την άλλη μα ζητάνε ε, να κάνουμε κάποιε επιλογέ, α πούμε. Κάποιε αξιολογικέ κρίσει. Εγώ δεν κάνω τώρα αξιολογική κρίση. Καταλαβαίνω τις ανησυχίε που υπάρχουν ε, για την απομόνωση μέσα στην οποία ζούμε ε, λόγω των προτιμήσεών μας, αυτό το filter bubble στο ίντερνετ. Ε, στο, βιβλιο, στο βιβλιοπωλείο όταν μπαίνουμε ας πούμε, ε, εμείς επιλέγουμε πραγματικά το βιβλίο μας. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το τι συμβαίνει στο ίντερνετ. Κάτι σε σχέση με αυτά που ο κύριος Μπλέτσας ε, Καταρχά πρέπει να διαχωρίσουμε τους διάφορους αλγόριθμους για να δούμε τι πρόβλημα έχει ο καθένας. Μπορεί να είναι διαφορετικά αυτά τα προβλήματα. Ακόμη και αλγόριθμοι για τα fake news μοιάζουν, πρέπει να τους διακρίνουμε. Έπειτα για τη διαφάνεια. Τουλάχιστον να μιλήσουμε για τις αρχές ε, πάνω στι οποίες θα εδράζονται οι αλγόριθμοι. Μιχάλη, η διαφάνεια είναι δευτερεύουσα ε, σε σχέση με την πρόθεση, με τη συζήτηση που θα κάνουμε για την πρόθεση του αλγορίθμου. Αν όλοι συμφωνήσουμε ως κοινωνία, ε, κλάδος, ε, κοινωνία των πολιτών, πολιτική κτλ. Ότι οι αλγόριθμοι οι οποίοι αφαιρούν τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι θετικό, μετά μπορούμε να μιλήσουμε το θέμα τη διαφάνεια και πώ θα το κάνουμε. Αλλά δεν έχουμε φτάσει στη φάση όπου έχουμε συμφωνήσει για το τι θα κάνουν ακριβώ, τι θα πρέπει να κάνουν οι αλγόριθμοι. Επομένω, η διαφάνεια είναι απαραίτητη, αλλά η συζήτηση για την πρόθεση και το τι πρέπει να ε, κάνουμε είναι σημαντικό και πρέπει να προηγηθεί. Για το παράδειγμα που ανέφερε ο κ. Χριστιανίνη για την εταιρεία Admiral. Ε, εμείς λέμε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε στοιχεία των ανθρώπων ας πούμε, για να ε, παίρνεις οικονομικές αποφάσεις. Οπότε τα κλείνουμε αυτά τα στοιχεία. Τα κοινωνικά μέσα δικτύωση ε, λένε, έχουν πολιτική που λένε δεν μπορεί να πάτε τα δεδομένα μου και να τα χρησιμοποιήσετε, α τα χρησιμοποιήσουν ας πούμε, οι ασφαλιστικέ εταιρείε κτλ. Και εσεί, α πούμε, όταν είσαστε μια εταιρεία ασφαλιστική, α πούμε, ε, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα στοιχεία. Δεν σα τα δίνουμε. Ακούσα πολλά ερωτήματα εδώ, με ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση σημερινή. Εγώ ε, εκπροσωπώ τον κλάδο, έτσι και αναγκαστικά. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή συμφωνήσουμε με την πρόθεση, ε, μετά μιλάμε για την διαφάνεια και μετά μπαίνουμε στη δράση. Γιατί η τεχνολογία κινείται πάρα πολύ γρήγορα και θα ε, ανησυχούσα βεβαίως αν οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα ας πούμε, δοθούν μόνο από την κυβέρνηση και όχι από την, τον κλάδο. Το βασικό είναι όμω να μην έρθουμε σε αντιπαράθεση εμεί, ο κλάδο δηλαδή και η κυβέρνηση. Το θέμα είναι να κάνουμε μια συζήτηση ε, επί τη αρχή. Um, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρίτσαρτ. Έχω μία ερώτηση να σου κάνω με βάση αυτά που είπε. Δηλαδή, μα είπε ότι οι πελάτε επιλέγουν τα βιβλία στο βιβλιοπωλείο. Αλλά υπάρχει εδώ ένα θέμα, ότι όταν πρόκειται για την αναζήτηση ε, που μιλάμε πρόκειται για ένα και μόνο βιβλιοπωλείο και το μεγάλο αφεντικό λέει ότι οι άνθρωποι ε, αναζητούν πληροφορίες και ελέγχουν με ποιον θα τις μοιραστούν, αλλά δεν μπορούν να πάνε σε άλλη πλατφόρμα. Ε, ποια είναι, ποιος είναι ο ανταγωνισμός ακριβώς εδώ. Σε τελική ανάλυση οι χρήστες εξαρτώνται από τους δικούς σας τους αλγορίθμους, γιατί εσείς είσαστε οι φρουροί. Πώς γίνεται ακριβώς το όλο θέμα με τον ανταγωνισμό. David, έχω να σου πω κάτι ευχάριστο. Έχουμε ένα συγκεκριμένο εργαλείο ε, μπορείτε να το κατεβάσετε και αυτό είναι ένα παράδειγμα ε, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Δηλαδή, ε, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν για τη φορητότητα, όμως υπάρχει αυτή η φορητότητα. Μπορεί κανείς όλες του τις πληροφορίες, όλα αυτά που έχει αποθηκεύσει, να τα μεταφέρει ε, μάλιστα αυτό υπάρχει εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια ακριβώς ε, και εμείς ε, διότι είμαστε επαφή με τους αρμόδιους που εκπονούν τους κανονισμούς. Άρα υπάρχει αυτό. Μετά, για τον ανταγωνισμό. λέγονται πάρα πολλά, αλλά εμείς και όλοι οι άλλοι που χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό από ό,τι υπήρχε ποτέ. Ε, οι άνθρωποι πλέον έχουν εξελιχθεί ε, και τα περισσότερα δεδομένα που χρειάζεται κανεί ε, είναι στο κινητό του, ακόμα και στο κινητό του. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα που βρίσκονται στο κινητό και οι χρήστες έχουν συνηθίσει να κατεβάζουν ένα app, να το κάνουν πολύ γρήγορα. Δηλαδή, οι χρήστες έχουν κάποιες επιφυλάξεις, αλλά όλοι έχουν καταλήξει στο ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να ενταχθεί κανείς σε ένα νέο κοινωνικό δίκτυο και με τον τρόπο αυτό οι αλγόριθμοι ελέγχουν και το τι ακριβώς υπάρχει στο κινητό σας και σε επαφές σας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε μελέτη περίπτωσης από δύο ανθρώπους που δουλεύουν σε διαφορετικούς, διαφορετικές θέσεις το χώρο της ενημέρωσης. Ο κύριος Γελάπης, ο οποίος ασχολείται με την τεχνολογία και ο συνάδελφός του ασχολούνται με την σύνταξη των ειδήσεων. Μπορούν να μας δείξουν πώς την πρακτική η τεχνολογία, πρακτικά η τεχνολογία πραγματικά μπορεί να έχει κάποια διαφορά. Καλησπέρα σας. Είμαστε οι τελευταίοι. Θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε λιγάκι, να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε και εμείς ε, τη ΣΤΟΑ που μας κάλεσε και θέλουμε να πούμε το εξής. Αυτά που βλέπετε είναι μια ιστορία για το πώς μπορούν να συνδυαστούν ένας μεγάλος φορέας και μία μικρομεσαία επιχείρηση για να φτιάξουν ένα τελικό προϊόν. Είναι μία επιτυχημένη ιστορία. Τα τρία T είναι η ομάδα, το team, με τα truth, η αλήθεια αυτή είναι μια πολύ σημαντική λέξη, δύσκολη στο χειρισμό της, αλλά θα σας ε, μιλήσουμε γι' αυτό. Και μετά το Τρούλι είναι ένα εργαλείο που έχουμε κατασκευάσει και τώρα έχει βγει και στην αγορά. Ξεκινάμε με το πρώτο τι; την ομάδα, το Team. ATC είναι μια μικρομεσαία στην Ελλάδα εδώ και 25 χρόνια και έχει δύο διαφορετικούς ε, κλάδους. Έχουμε ένα εργαστήρι καινοτομίας, ε, προσφέρουμε νέες ιδέες, ε, έχουμε πάρα πολλά πολλά έργα που μας αναθέτει η Κομισιόν, αλλά έχουμε και παραγγελίες από τη Silicon Valley. Και γι' αυτό σήμερα είμαστε σε πολύ καλή θέση. Στα προϊόντα μας, μόλις τα φτιάξουμε, τα, διαδίδουμε, τα πουλάμε σε 5 ή 10 χώρες και μετά συστήνονται ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Εμείς ασχολούμεθα περισσότερο με τα μέσα ενημέρωσης. Ε, συσταθήκαμε ε, κατά διάρκεια των Ολυμπιακών Αγών. Από τότε ε, προσφέρουμε συστήματα ενημέρωσης για ειδησιογραφικά δίκτυα, για εκδότες να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και επίσης προσφέρουμε και εφαρμογές για εταιρικές επικοινωνίες. Άρα δηλαδή εργαζόμαστε στενά με δημοσιογράφους. Πάμε στο άλλο τι, το truthness, ε, την ειλικρίνεια. Έγινε μια σχετική ενημέρωση στη Βουδαπέστη πριν από δύο εβδομάδες επ' αυτού. Και πάμε στην Deutsche που όλοι τη γνωρίζουν. Εγώ είμαι ο Βίλφχετ Χούντε από την Deutsche Welle. Χαίρομαι που είσαστε ακόμα εδώ. και θα έλεγαν να μείνετε, να μας ακούσετε, γιατί αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι ε, να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα, όχι τόσο για το μέλλον, όσο για το παρόν ίσως και για το παρελθόν. Εγώ εκπροσωπώ την Deutsche Welle. Ραδιοτηλεοπτικό σταθμό στη Γερμανία, ασχολείται με διεθνή θέματα. Ε, συνεργαζόμαστε με 60 περίπου χώρες, ε, προσφέρουμε ειδήσει σε πάρα πολλές γλώσσες και επίσης εμείς ε, προσφέρουμε ειδήσει ε, για όλες τις πλατφόρμες. Μπορείτε να μας βρείτε και ε, σε αυτά τα, τις μικρές συσκευές. Ε, βλέπετε λοιπόν εδώ Μερικές φορές η ελληνογερμανική συνεργασία μπορεί να είναι πολύ επιτυχημένη. Βλέπουμε και στη διαφάνεια. Κύριος Ζαγοράκης, τον βλέπετε εδώ, Τώρα είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βεβαίως δεξιά είναι ο κύριος Ρεχάγκελ, ο Ρεχάκλης όπως τον λένε στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στην, ε, στα δυσάρεστα. Αυτό που θα δείτε είναι το 2% μιας παρουσίασης που κάνω συνήθως, Λάλα Πένσεν Φάρα, and Fire. Αυτή είναι συνήθως η ομιλία που κάνω. Ε, και αφορά ε, τον χώρο της ε, ενημέρωσης. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα παράδειγμα. Πριν από ένα χρόνο προέκυψε αυτό, όπου διαπιστώσαμε ότι χρειάζονται δύο μόνο tweet για να προκύψει πυρηνική απειλή. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν που πίστεψε ένα ψεύτικο tweet και απείλησε με πυρηνική επίθεση. Άρα δηλαδή σήμερα που αυτό μπορεί να συμβεί με δύο μόνο tweet, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ε, και αυτοί που πρέπει να το αντιμετωπίσουν είναι όλοι αυτοί που κάθονται εδώ στο πάνελ, που μας μίλησαν. Επίσης όμως και οι δημοσιογράφοι, τα ειδησιογραφικά πρακτορία, τα γραφεία ειδήσεων. Ας δούμε τι συμβαίνει σε αυτά τα γραφεία ε, ή τι συνέβη κατά το παρελθόν με όλα αυτά που συνέβησαν. Και επειδή είμαστε στις Βρυξέλλες, ας ξεκινήσουμε με ένα πράγμα που είναι στάνταρτ για ειδησιογραφικά πρακτορία σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιούν εικόνες από αρχείο και υποτίθεται τις προσβάλλουν ως επίκαιρες. Αυτό εδώ το κλιπ, <laughs> θα βλέπετε, το είδα σε πάρα πολλά σημαντικά δίκτυα μία συγκεκριμένη μέρα και δεν θέλω να ξαναγίνει αυτό. Ε, και άλλα παραδείγματα από τις ε, βόμβες που είχαμε την επίθεση στο Μάντσεστερ. Βλέπετε τι συνέβη, συνέβη αυτό που όλοι γνωρίζουμε, τα tweet και εδώ ένα tweet που λέει ότι ένας γκάνγκστερ έξω από ένα νοσοκομείο αυτό αναπαρήχθη πάρα πολλές φορές, υπερβολικά πολύ και μετά κάποια μέσα ενημέρωσης και έχω συγκεκριμένα παραδείγματα, αρκετά μέσα ενημέρωσης το πίστεψαν και το μετέδωσαν με τον τρόπο αυτό αυτή η ψευτική είδηση ε, αναπαρήχθη και γι' αυτό έπρεπε να παρέμβει η αστυνομία και να το διορθώσει. Φαύλος κύκλος δηλαδή. Θα θυμάστε αριστερά, Las Vegas, πρόσφατα, αυτόν που βλέπετε κάτω από το Breaking News αυτός ε, κατηγορείται άδικα ότι δίθεν αυτός ο άνθρωπος διέπραξε όλα αυτά τα ειδεχθή εγκλήματα. Λάθος. Και θα σας δείξω στο τέλος της ομιλίας μου πώς το ανακαλύψαμε και άλλοι βέβαια. Θέλω απλά να σας ε, δείξω το πόσο περίεργο και παράδοξα είναι αυτά που συμβαίνουν. Εδώ βλέπουμε ένας Γερμανός ε, ποδοσφαιριστής που και αυτός υποτίθεται ότι ήταν ε, αγνοούμενος σε αυτή την επίθεση. Λάθος και αυτό. Αλγόριθμοι κάνουν πολύ καλή δουλειά, αλλά οι αλγόριθμοι κάνουν και λάθη, λάθος πράγματα. Ακούσαμε, ε, τέθη ένα ερώτημα ε, και απαντήθηκε ότι και στις μηχανές υπάρχει ένα ποσοστό λάθος. Λυπάμαι ε, που δείχνω όλα από την Google που είναι λάθος, έχω όμως και άλλα από το Facebook, μην ταράζεστε από την Google. Μία θεωρία συνωμοσίας που προέκυψε από μια θεωρια συνωμοσια που προκατηλημένη πηγή και τελειώνει την ε, ιστορία ε, εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα με πάρα πολλές λάθος ειδήσει που ε, μεταδόθηκαν σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό δεν επιτρέπεται, δεν πρέπει να συμβαίνει, διότι η δημοσιογραφία και αυτή είναι, αυτός είναι ο ορισμός του Καρλ Μπέρνστιν, ο οποίος αποκάλυψε το σκάνδαλο του Watergate, ο οποίος είπε ότι η δημοσιογραφία είναι η βέλτιστη, εφικτή εκδοχή της αλήθειας. Αλήθεια όμως τι είναι, υπάρχει μόνο μία αλήθεια σήμερα. Για τους δημοσιογράφους τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα από ποτέ το να βρουν αυτήν την αλήθεια για να μπορούν να παράγουν ένα συγκεκριμένο προϊόν και οι δημοσιογράφοι έχουν εργαλεία, έχουν ε, τους υπολογιστές, ε, μπορούν να γυρίσουν βίντεο, ε, να φτιάξουν ιστοσελίδες, αλλά δεν έχουν αρκετά εργαλεία για να μπορούν να στηρίξουν τη διαδικασία επαλήθευσης. Και Γιάννη, τώρα εσύ, να τη φτιάξαμε εμείς. Θα πω δύο λόγια για την απαρχή αυτής της ιδέας, από πού ξεκινήσαμε. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ την ε, Κομισιόν γιατί ήταν πρωτοπόρος το 2010-2011. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Το πρόβλημα δεν ήταν τόσο έντονο όπως σήμερα. Ε, δεν ήταν κάτι που μας απασχολούσε στην καθημερινότητά μας. Ξεκινήσαμε με έναν ε, σένσορα, κοινωνικό σένσορα, ένα ε, πρόγραμμα που εστίαζε στην έρευνα και το πώς θα εξάγουμε πληροφορίες. Συνεχεία. Πήγαμε στο Reveal που ήταν ένα πρόγραμμα επαλήθευσης. Ε, ήρθαμε σε επαφή με τις μεγαλύτερες οργανώσεις στην Ευρώπη ε, και είδαμε τι κάνουν χειρονακτικά, γιατί έχουν μεγάλες ομάδες που κάνουν επαληθεύσεις. Και το, αυτό το συνδυάζουμε με την τεχνητή νοημοσύνη για να εκπαιδεύσουμε το, το μηχάνημά μας. Και επίση ε, φτιάξαμε και μια συνεργατική πλατφόρμα, ούτω ώστε να συνεργάζονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, δεν χρειάζεται να είναι σε μια συγκεκριμένη χώρα, για να αξιολογούν μαζί, να κρίνουν μαζί. Α πάμε και στη δομή τώρα. Τα τρία project που έχουμε είναι τα τρία στατικά. Είναι το συνολικό τα συνολικό περιεχόμενο που βρίσκει από τι διάφορε πηγέ κοινωνική δικτύωση και συλλέγει πραγματικά δεδομένα, μετά οργάνωση, οργανώνει αυτά τα δεδομένα και δουλεύεις σαν ομάδα και εσωτερικά αλλά και με εξωτερικού ε, ε, εμπειρογνώμονες και το τρίτο τμήμα είναι η επαλήθευση. Χρησιμοποιεί ε, εργαλεία από τρίτου για επαλήθευση αλλά και όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι μεγάλοι οργανισμοί που, γίνονται, που κάνουν αυτόματη επαλήθευση. Θα πάω τώρα στο Truly Media. Εδώ έχουμε λίγα παραδείγματα, αλλά είναι πραγματικά από τις μέρες που έγιναν και τότε είχαμε αυτές τις εικόνες για να καταλάβετε που το Truly υποστηρίζει ε, την διαδικασία επαλήθευσης και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και αλγόριθμοι εν δράση, είδαμε τι βλέπουν οι δημοσιογράφοι για να πάρουν τι αποφάσει του. Βλέπετε αυτή τη φωτογραφία, υπήρχε στο Twitter, βλέπετε το λογαριασμό. Τι σα δίνει η πλατφόρμα την πρώτη στιγμή, σα δίνει ε, αυτή την εικόνα από το truthness, από το μοντέλο truthness και την δραστηριότητα αυτή τη πηγή και κάνει και κάποιε διασταυρώσει. Ε, ε με γνωστέ πηγέ παραπληροφόρηση, ε, τι κοιτάνε οι δημοσιογράφοι, ίσω τι κοιτάνε για πρώτη φορά και λένε Α, ύποπτο λογαριασμό. Αυτό το άτομο είναι σε ένα κατάλογο που δεν, ε, μη αξιόπιστων πηγών. Το λαμβάνω υπόψη στην διαδικασία επαληθευσή μου. Το ίδιο και εδώ. Βλέπετε τα πραγματικά αποτελέσματα. Αυτόματα γίνεται σε μία διεπαφή. Μιλάμε για αλγόριθμους και για API. Ε, για το Truthness διερωτάμε διάφορους στην Google ε, και παίρνουμε τα αποτελέσματα και δίνουμε ε, στοιχεία ε, πάρα αυτά στους δημοσιογράφους για διαδικασία επαλήθευσης. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, πρέπει, κοιτάμε τη χρονική στιγμή ε, που έγινε ο ισχυρισμός και βλέπουμε ότι δεν είναι η πραγματική πρωτότυπη εικόνα. Ε, δεν είναι εικόνα από τη στιγμή που έγινε αυτό το γεγονός, αλλά αναρτήθηκε πολύ αργότερα. Ε, όλα αυτά τα στοιχεία τα λάβουν υπόψη οι δημοσιογράφοι να πάρουν την απόφαση. Και να το Κολοράντο εδώ τελευταία Κάτι που σας διέφυγε ίσως ε, Εδώ ακούμε, φανταστείτε, σε διάφορες γλώσσες διάφορους ισχυρισμούς. Ίσως δεν ήταν στα, στους πηχαίους στην ε, Ευρώπη. Ε, ήταν ένας πυροβολισμός υποτίθεται στο Κολοράντο. Είδαμε αυτή την είδηση, λέμε, αυτό το άτομο είναι καλά συνδεδεμένο, έχει καλή φήμη στο Twitter. Θα μπορούσαμε να επαληθεύσουμε επίσης μαζί με την Google και να διασταυρώσουμε με χάρτες της ε, Google για να δούμε πότε ε, πήρε κανείς αυτή την εικόνα, αυτή τη φωτογραφία. Πού ήταν κοντά και η αξιολόγηση του δημοσιογράφου είναι επαληθεύτηκε αυτό το στοιχείο, μπορώ να τη, να χρησιμοποιήσω αυτή την είδηση. Όμως με, όλες αυτές, με όλα αυτά τα στοιχεία από την ε, τεχνητή νοημοσύνη, μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για μια πλατφόρμα συνεργατική. Μπορεί να καλέσει φίλου σου, ανθρώπου από άλλε οργανώσει για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επαλήθευση. Ε, Επίση, ε, έχουμε πληροφορίε καιρού, ε, διάφορα στοιχεία, ας πούμε, από ιατροδικαστές. Όλα αυτά είναι στοιχεία που τα βάζουμε μέσα στο σύστημα. Τα επόμενα βήματα. Ε, μετά τις γενικές, ε, γερμανικές εκλογές πήγαμε στο beta testing. Εκεί συμμετείχε και η Deutsche Welle. Έχουμε περάσει στην εμπορική εκδοχή. Επίσης υπάρχει μια μικρή θυγατρική εταιρεία, ένα η πρώτη, ο πρώτο πελάτη είναι το MIT και η Deutsche Welle και εγώ κάθομαι <laughs> ανάμεσα στου δύο. Είναι οι καλύτεροι πελάτες μας. Και κάτι νέο, κάτι καινούριο. Τελευταία νέα. Και, μια, και είναι τα τελευταία νέα θα πρέπει να τα πει ο συνάδελφος που μιλάει για νέα, για ειδήσει. Στο τέλος μιας παρουσίασης ε, πάντα υπάρχει και κάτι ακόμα. Έχουμε και εδώ κάτι ακόμα, όπως είπε ο Γιάννης. Το μάθαμε σήμερα το πρωί, αυτό το έξτρα πράγμα. Και είτε θα έχουμε την αποκλειστικότητα, και δεν το λέω για πλάκα, είναι η πρώτη φορά που το λέμε δημόσια. Η πρώτη σύμβαση και ο πρώτος πελάτης που θα πληρώσει για το Truly Media είναι η Διεθνής Αμνηστία. Η Διεθνής Αμνηστία που δεν μην σας ε, φαίνεται για εταιρεία ΜΜΕ, αλλά αυτό που κάνει με τη θαυμάσια δουλειά της είναι να ψάχνει, να επαληθεύει και να τεκμηριώνει όλα τα είδη παραπληροφόρησης και φρικαλαιοτήτων ανά τον κόσμο. Και θα χρησιμοποιήσει το προϊόν μας, το Truly Media, μετά από μια σύντομη μεταβατική περίοδο, στις αρχές του 2018. Από εκεί θα ξεκινήσει και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη συνεργασία. Αυτά, ευχαριστώ. Thank you, Giannis, uh, and thank you, Wilfred. You can always... Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Και ξέρετε, οι δημοσιογράφοι θέλουν ε, να έχουν πάντα μια αποκλειστική είδηση. Μπορείτε να τους το πείτε αυτό, αυτή την είδηση. Εγώ πάντως ε, βλέπω ότι όλα αυτά διαδίδονται σε πάρα πολλά γραφεία που ασχολούνται με ειδήσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Πριν λοιπόν περάσουμε σε ερωταπαντήσεις, ε, φαντάζομαι ότι θα θέλετε να κάνετε ουσιαστικές ερωτήσεις, όχι τοποθετήσεις ή ομιλίες. σύντομα, τρία λεπτά μόνο. Ε, θα μας μιλήσει ο κύριος ε, Τσεζάρη, ο οποίος ε, είναι από την DG Connect, η Γενική Διεύθυνση Connect και θα μιλήσει για το project σχετικά με τις ψευδείς ειδήσει. Δεν θέλω να αφαιρέσω χρόνο από τη συζήτηση, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΣΤΟΑ για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, πολύ χρήσιμα αυτά που ακούσαμε για την δουλειά που θα έχει να αντιμετωπίσει και η Κομισιόν, η οποία όπως γνωρίζετε ανακοίνωσε τη Δευτέρα μία πρωτοβουλία μετά από ένα αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και μετά από ένα ψήφισμα του Ιουνίου, η Κομισιόν σκέφτηκε ότι θα πρέπει σιγά σιγά να δει τι θα κάνει ε, σχετικά με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, ε, επιγραμμικά κυρίως. Αυτά που ακούσαμε σήμερα, τα τεχνικά κυρίως, είναι πολύ χρήσιμα για τη δουλειά μας στο μέλλον. Και αυτά που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να οργανώσει ε, διαρθρωμένο διάλογο με όλους τους ε, άμεσα ενδιαφερόμενους που εκπροσωπήθηκαν πολύ καλά σήμερα. Οι πλατφόρμες, τα μέσα ενημέρωσης, οι ερευνητές και θέλουμε και επικοινωνία με τις ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, γιατί είναι εκείνοι οι οποίοι διαπιστώνουν ε, τις επιπτώσεις στην κοινωνία. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτές οι οργανώσεις να ενταχθούν στο διάλογο. Το τελευταίο που θέλω να πω αφορά σε κάποια τεχνική φύσεω θέματα. Ε, τα βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Νομίζω ο βασικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή είναι να κατανοήσουμε καλύτερα την ποικιλομορφία των ε, πληροφοριών, την αξιοπιστία αλλά και τη διαφάνεια του ίδιου του συστήματος και όσον αφορά την ροή χρηματοδότησης που απευθύνεται στην ενημέρωση. Όσον αφορά αυτή την ποικιλομορφία, άκουσα πολλά και ενδιαφέροντα. Ότι δηλαδή θα πρέπει να διαφοροποιούμε ανάμεσα στους διάφορους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται. Είναι αυτοί που έχουν το περιεχόμενο, έχουμε αλγορίθμους που ε, οργανώνουν το επιγραμμικό περιεχόμενο και αυτοί εξελίσσονται, αναπτύσσονται περαιτέρω. Νομίζω ότι πρέπει να εξελιχθούν περαιτέρω τα εργαλεία και υπάρχει κάποιος συσχετισμός ανάμεσα ε, στις ε, ψευδείς ειδήσει και την πόλωση και σχέση ανάμεσα στην πόλωση και τα filter bubbles και τα eco chambers. Ε, έχουμε λοιπόν πάρα πολλά που μοιάζουν και ίσως αυτή να είναι η ρίζα του προβλήματος. Άρα, εφόσον θέλουμε διαφοροποίηση, πρέπει να έχουμε και διαφοροποίηση σε αυτά που δίδουμε στους χρήστες μέσα από τις πλατφόρμες. Αυτό είναι καθοριστική σημασία. Ο αγώνας για την αλήθεια είναι ο αγώνας για ένα σύστημα όπου μειώνεται το επίπεδο της πόλωσης και κυρίως σε εκείνα τα θέματα όπου ε, υπάρχει μία τάση συγκέντρωσης και αυτό αφορά όχι μόνο προεκλογικές εκστρατείες αλλά αφορά και τομείς όπως είναι η υγεία, το περιβάλλον, η οικονομία, η μετανάστευση. αυτή είναι τομείς όπου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και τέλος, νομίζω το παράδειγμα που αναφέρθηκε μόλις τώρα είναι χαρακτηριστικό ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα σε σχέση με τον έλεγχο των γεγονότων. Καλά αυτά που γίνονται, αλλά θα πρέπει να συμβαδίζουν και με μια επιπρόσθετη προσέγγιση που θα επιτρέπει τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. Αλλιώς απλά θα εντοπίζουμε ζημιά που έχει ήδη γίνει. Αυτό ελπίζω ε, να έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε κυρίως σε επίπεδο ομάδας υψηλού επίπεδου που έχει συστήσει η Επιτροπή και που θα αρχίσει την, ε, τις εργασίες της τον Ιανουάριο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάολο για την παρέμβασή του και τώρα έχουμε χρόνο για ερωταπαντήσεις. Να μας ε, συστήνεστε πρώτα και παρακαλώ. Ο κύριος ε, Πάολ Ρούμπικ από τη ΣΤΟΑ, την Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική για μας και όλοι βεβαίως έχουμε αυτές τις νέες συσκευές. Το κινητό του δείχνει ο κύριος ε, Ρούμπιχ. Ξέρουμε τι διαβάζουμε, αλλά δεν ξέρουμε από πού προέρχονται οι πληροφορίες στα κινητά. Και δεν γνωρίζουμε επίσης ποιος έχει πρόσβαση στα κινητά μας. Μήπως γνωρίζετε κάποιες ε, τεχνικές επιστημονικές δυνατότητες για να μπορούμε να εντοπίσουμε ποια app συνδέονται με ποια app, ποιος έχει πρόσβαση στις συσκευές μας και όταν κατεβάζει κανείς ένα app είναι απαραίτητο να συμφωνεί και να αποδέχεται τα cookies που προτείνουν. Ε, Πώς μπορεί κανείς να διαφυλάξει την διαφάνεια και την ιδιωτικότητα. Ήμουνα ε, πρόσφατα στο MIT και εκεί γνώρισα έναν καθηγητή με τη δική του ομάδα που προσπαθούν να αναλύσουν τι συμβαίνει στο παρασκήνιο. Πιστεύετε ότι υπάρχει υπάρχουν δυνατότητες να γνωρίζουμε καλύτερα ε, πού ε, κατευθύνονται τα δεδομένα και μπορούμε να τα αναχαιτήσουμε χωρίς να διατρέχουμε κίνδυνο να βρεθούμε τελικά και χωρίς ε, συσκευή. Μπορείτε να μας απαντήσετε αν υπάρχει αυτή η σχετική τεχνολογία και πώς μπορούν να απαντηθούν τα ερωτήματα περί διαφάνειας. Ε, κοιτάξτε, θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα να ε, χαρτογραφηθούν όλα τα app και πώς συνδέονται μεταξύ τους. Το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν έχουμε σαφείς κανόνες. Δεν έχουμε σαφείς κανόνες για το σε ποιον θα δίνουμε την άδεια. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο βελτίωσης και υπάρχει και μεγάλο περιθώριο βελτίωση όταν αφορά, όσον αφορά τα metadata. Αν δείτε τις ε, έρευνες σχετικά με τον έλεγχο των γεγονότων, την αλήθεια, έλεγχο αλήθεια στα μέσα ενημέρωσης, θα διαπιστώσετε ότι τα περισσότερα γίνονται στο Twitter. Και ο λόγος που γίνονται στο Twitter είναι ότι για κάθε tweet παρά το γεγονός ότι βλέπουμε μόνο 140 χαρακτήρες, μιλάμε για 5K, δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερο γιατί, διότι υπάρχουν τα metadata τα οποία μας επιτρέπουν να ε, ιχνηλατούμε τη ροή των πληροφοριών. Πράγματι, χρειαζόμαστε ε, χαρτογράφηση, αλλά χρειαζόμαστε και συσκευές ιχνηλάτησης. Τα metadata μας δίνουν αυτή την ευκαιρία, μας επιτρέπουν την ανάλυση με μεγαλύτερη διαφάνεια. Και νομίζω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι Σήμερα μιλήσαμε για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ε, αυτοί που προβλέπουν με ακρίβεια και ελέγχουν την ακρίβεια ε, της αλήθειας σε ένα tweet, αυτό έχει σχέση με την προέλευση. Συνήθως ε, οι μη επαληθευμένες ειδήσει ε, έχουν την ίδια πηγή, όταν έχουμε επαλήθευση έχουμε πολλές πηγές. Οι άνθρωποι κάνουν tweet πάνω στο tweet. Άρα δηλαδή αν κάτι απαντηθεί με tweet από κάποιον ο οποίος έχει ε, πολλούς ε, follower ε, και απαντάει σε κάποιον που έχει όμως λίγους follower, αυτό πιστοποιεί μάλλον την αλήθεια. Και το αντίθετο την ψευδή είδηση. Έχει δηλαδή κανείς κάτι τέτοια τρίκ, άρα χρειαζόμαστε και χαρτογράφηση, αλλά χρειαζόμαστε και σαφέστερους κανόνες για τα metadata. Και νομίζω αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία ε, για τις υπόλοιπες πλατφόρμες ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Twitter. Διδιέ Κανέ λέγομαι. Είμαι Βέλγος. Ένα από τα προβλήματα για τις ψευδείς ειδήσει και τις αληθείς ειδήσει είναι ότι οι ψευδείς ειδήσει ε, συνήθως είναι δωρεάν. Ενώ για τις αληθινές ειδήσει πρέπει να πληρώσεις, πρέπει να πας στο Elsiv ή αλλού. Ας πούμε, θα μπορούσα να δώσω και άλλα παραδείγματα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ε, πολεμούν να έχουμε επιστημονικά δεδομένα ε, που ειδικά όταν αυτά προκύπτουν από δημόσια χρηματοδότηση τουλάχιστον να είναι διαθέσιμα, προσπελάσιμα στο διαδίκτυο. Κύριε Κλιάφα, ε, τι πιστεύετε. Οι επιστημονικές πληροφορίες που τις παράγουμε πληρώντας με δημόσιο χρήμα δεν θα έπρεπε να είναι κάτι που είναι δωρεάν στο διαδίκτυο, δεν θα πρέπει να το ξαναπληρώσουμε. Επίσης, κανένας δεν μιλήσει σήμερα για την Wikipedia και για την ελεύθερη πληροφορία που υπάρχει εκεί. Τι θα μπορούσατε να μου πείτε γι' αυτό. Θέλετε να μιλήσετε εσείς. Ε, ή και ο άλλος ε, κύριος, ο κύριος Βλάχος, ας πούμε, μπορεί να, και αυτός να συμμετάσχει, αν θα πρέπει οι, αυτές οι πληροφορίες να υπάρχουν δωρεάν. Δεν μου απευθύνθηκε η ερώτηση, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχουν δημόσια μέσα ενημέρωσης. Αυτή είναι η δωρεάν εναλλακτική για ποιοτικό, ποιοτική δημοσιογραφία. Το BBC, Deutsche Welle και άλλοι εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι πλεονέκτημα του πλουραλισμού των ΙΜΕ εδώ στην Ευρώπη. Εσείς βεβαίως αναφερθήκατε σε επιστημονικό περιεχόμενο και τα αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων. Ε, από την εμπειρία που έχουμε από ερευνητικά προγράμματα, ε, ξέρουμε ότι υπάρχει υποχρέωση και υπάρχει και στη σύμβαση. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας πούμε, υποχρεώνει τις εταιρείε να, να δημοσιεύουν σε, μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα το προϊόν τους. Ε, και αυτό είναι θετικό. Κόλμαν. Θα κάνω μια διάκριση ανάμεσα στην ποιοτική πληροφόρηση και αυτό που αναφερθήκατε σε, ως ψευδείς ειδήσει. Για να έχετε ποιοτική πληροφόρηση χρειάζεστε ε, ένα μοντέλο για να διατηρήσετε το υψηλό επίπεδο. Εγώ είμαι υποστηριχτής ε, της ανοιχτής πρόσβασης ε, που όμως δεν είναι δωρεάν. Κάποιος πρέπει να υποστηρίξει, να χρηματοδοτήσει αυτή την ανοιχτή πρόσβαση. Το κάνουν οι εκδότες. Οποιοςδήποτε θέλει ανοιχτή πρόσβαση ε, και θέλει να, έχει, να συμμετάσχουν μεγάλοι εκδότες στο Elsevier, ε, είναι θαυμάσιο μοντέλο και είναι στη διάθεση όλων των πολιτών. Παρακαλώ, η κυρία. Ε, thank you very much. Um, Ευχαριστώ. Χάνα Μαριτήλο. Γερμανίδα είμαι. Μία ερώτηση για τον ε, έλεγχο των ε, δεδομένων. Ε, αυτό είναι το ανάχωμα εναντίον των fake news. Ε, όμως δεν υποσκάπτουμε έτσι την, το, το την τέταρτη εξουσία ε, που ότι θα έπρεπε να κάνουν αυτοί αυτόν τον έλεγχο. Ενώ τώρα οι, κάποιοι ανεξάρτητοι άνθρωποι, κάποιοι που δεν έχουν σχέση με τον τύπο, ας πούμε, ελέγχουν τους ελεγκτές, ας πούμε. Και τι θα γίνει ε, αν κάποιο ελεγχει ελέγχει, κάνει fact-checking, δηλαδή αυτόματα ας πούμε, ε, κάποιου πράγματος το οποίο έχει ελεγχθεί ήδη. Τελικά το θέμα αυτό ε, καταλήγει στο ζήτημα της διαφάνειας. Έχετε δίκιο. Η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική. Ε, ο έλεγχο των δεδομένων, αυτόματο ή όχι, και οι δύο θα πρέπει να έχουν ένα δεύτερο επίπεδο ελέγχου και να υπάρχει και λογοδοσία για όποια λάθη. Συμφωνώ με εσά και με το, τη δήλωσή σα με την ανθρώπινη, τον ανθρώπινο έλεγχο έχουμε μία έκθεση, όχι απλώς ένα αποτέλεσμα σωστό ή λάθος, όχι πάντα βέβαια, αλλά με τους αλγόριθμους τα πράγματα μπερδεύονται. Γιατί προσπαθούμε ακόμα να μάθουμε και να ερμηνεύσουμε τους αλγόριθμους. Είτε λόγω σχεδίου, είτε γιατί έχουμε ένα μοντέλο και να ερμηνεύσουμε το μοντέλο, υπάρχουν πάρα πολλά, πολύ φαύλοι κύκλοι και πολλά καυτά θέματα γύρω από αυτό το ζήτημα των αλγορίθμων. Σας κάλυψα. Εμείς ε, στη Facebook ε, προσπαθούμε να συνεργαστούμε με αυτούς που ελέγχουν τα γεγονότα και τα πράγματα είναι περίπλοκα. Και υπάρχει το εξή. Υπάρχουν ε, οργανώσεις, εταιρείε που κάνουν αυτό τον έλεγχο των γεγονότων. Και το θέμα είναι τι κάνουμε. Δηλαδή ζητάμε από έναν φορέα να ελέγξει έναν άλλο. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Κατόπιν, σε πάρα πολλές χώρες ο έλεγχος των γεγονότων γίνεται, είναι κάτι που η αριστερά κάνει προς τη δεξιά. Δηλαδή η μία πλευρά ελέγχει την άλλη. Παράδειγμα το Brexit. Το να βρει κανείς ε, πραγματικά ουδέτερους ελεγκτές των γεγονότων, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και επίσης είναι και πολύ δύσκολο να γίνεται έλεγχος και να υπάρχει και η αντίθετη πλευρά του άρθρου, αλλά ε, το θέμα είναι ότι πράγματι ε, θα πρέπει να εμφανίζεται ένα άρθρο και όλοι να γνωρίζουν ότι μετά έχει γίνει έλεγχος ουδέτερος. Πιστεύω όμως ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορεί να γίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι εδώ ε, υπάρχει μια επανάσταση. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν είχαμε αρκετές πληροφορίες, ε, νομίζω υπάρχουν αρκετά ωφέλη, ε, υπάρχουν πολλές πληροφορίες, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Και ο έλεγχος των γεγονότων και οι αρχές της επιστημονικής μεθόδου πρέπει να διδαχθούν ε, στα σχολεία. Ίσως τώρα πράγματα δεν κάνουμε πολύ καλή δουλειά από αυτού. Είμαι ο Βαλεντίνος από την Ελλάδα. Ερώτηση προς τον Άλαν από το Facebook. Όπως είπατε, το Facebook ε, προσπαθεί να αντιμετωπίσει κακή συμπεριφορά και fake news. Το πρόβλημα είναι ότι προσπαθείτε συνεχώς να αντιμετωπίσετε ε, το τι γίνεται τώρα αλλά δεν προσπαθείτε για το μέλλον να εκπαιδεύσετε τους χρήστες, να τους ε, παρουσιάζετε άλλες απόψεις και να υπάρχει κάποια έτσι κριτική με κάποια μια άποψη με κριτική. Δηλαδή όλοι λένε τα fake news είναι πρόβλημα, όλοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα fake news ε, τεχνικά και τεχνολογικά, αλλά κανείς δεν το πράττει σε ανθρώπινη βάση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ξέρετε, στο τέλος του 2016 ε, όλοι ε, συνειδητοποίησαν το τι συμβαίνει και εταιρείε σαν τη δικιά μας ε, ανέλαβαν διάφορες πρωτοβουλίες. Εμείς κάναμε και το εξής. Καταβάλαμε, πληρώσαμε για ολοσέλιδες καταχωρήσεις ε, στις εφημερίδες σχετικά με το πώς πρέπει κανείς ε, να ενημερώνεται για τα μέσα ενημέρωσης. Ε, δηλαδή, μία εκπαίδευση, αν θέλετε, για τα μέσα ενημέρωσης. Η εκπαίδευση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν μπορέσει κανείς να το αντιμετωπίσει, κατά κάποιο τρόπο έχει αντιμετωπίσει και το πρόβλημα συστημικά δηλαδή οι άνθρωποι να κατανοούν ε, τις ε, πηγές ε, και αν το κάνει κανείς αυτό δεν θα χρειαστεί να επεμβαίνει ο ίδιος στις πηγές. Ας πούμε το να πει κανείς ότι ο εμβολιασμός είναι επικίνδυνος, αυτό θα έπρεπε να μπορεί κανείς να το ελέγχει χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει σε άλλα τρίκ με οικογένειες και το καθεξής. Και πάλι σας λέω, ε, δαπανίσαμε χρήματα για καταχωρήσεις εφημερίδες, ε, πρωτοφανές αυτό για μας ε, και θα το κάνουμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς τον κύριο Κριστιανίνη. Συμφωνείτε ότι η σημερινή κατάσταση, η διοντολογική κατάσταση του Facebook είναι ε, μέσω της αυτοδιόρθωσης. Ε, υπάρχει δηλαδή ένας βρόχος ανατροφοδότησης. Το λέω γιατί ο κύριος Μοέδας μίλησε για την τιμωρία, για την περίπτωση παραβίασης του κώδικα διοντολογίας. Γιατί είμαστε τόσο ανεκτικοί. Ήμασταν τόσο ανεκτικοί μέχρι τώρα. Είναι γιατί η πρόοδος είναι τόσο τρομακτική, ας πούμε, που πρέπει να... που μπορούμε να δεχτούμε κάποιες ζημιές στην κοινωνία. Ε, η προέλευση της λέξης ε, διοντολογία, ethics, είναι στο, βασίζεται στην ελληνική λέξη ήθος. Ε, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για αυτό το θέμα. Um, I σας βλέπω για να σας απαντήσω. Αυτό το θέμα δεν θα το ρυθμίσουμε με, το, με τους αλγόριθμους. Το θέμα τελικά είναι θέμα αξιών. Και οι αξίες ε, μετατρέπονται, αλλάζουν ε, με πολύ αργούς ρυθμούς. Το ήθος, το έθος αλλάζει πάρα πολύ αργά. Ε, η τεχνολογία όμως πάρα πολύ γρήγορα. Προσπαθούμε λοιπόν να, να τα φέρουμε σε φάση. Ρωτάτε αν υπάρχει ένα σύστημα ανατροφόδησης. Αυτό που έχω να σας πω στις προηγούμενες επαναστάσεις, την Αγγλική Βιομηχανική Επανάσταση, ήταν ένα ε, τεχνικό, μια τεχνικό μηχάνημα, η ατμομηχανία, ας πούμε, που οδήγησε σε διάφορες ε, αλλαγές, που οδήγησε σε, στο σοσιαλιστικό κόμμα, στα, στα, σχολεία, τα πάντα, ας πούμε, ξεκίνησαν με αυτό το μικρό, ας πούμε, ε, φαινόμενο. Εκείνη την εποχή ε, δεν μπορούσε να το αποφύγεις αυτό. Και εμείς ε, μπορούμε να δεχτούμε ότι ισχύει αυτή η αναλογία. Ε, θα αλλάξουν τα πάντα. Τα έθιμά μας, η πολιτική μας. Το θέμα είναι, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση χωρίς να περάσουμε από τον πόνο και την οδύνη της βιομηχανικής επανάστασης. Βλέπουμε ότι αλλάζουν οι αξίες από γενιά σε γενιά και διαμορφώνουν και τις κοινωνίε μας. Θα ακούσουμε τις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Ο κύριος. Είμαι από την Ολλανδία σύμβουλος. Όταν άκουσα ε, τον κύριο από την Google ανησύχησα όταν μας είπατε ότι κάποιες πληροφορίες τις φιλτράρετε ε, Δηλαδή σας προσφέρετε η δυνατότητα να φιλτράρετε πληροφορίες. Αυτό κατ' ουσίαν όμως είναι λογοκρισία. Εντάξει, για το ο, ολοκάπτωμα, φρικτά αυτά, ε, αυτά όμως είναι λογοκρισία και έχουν και σχέση και με ε, την ανάληψη ευθυνών. Δηλαδή μπορεί κανείς... Ε, να αναλάβει αυτό το έργο της λογοκρισίας ή μήπως αυτό θα πρέπει να γίνεται ανάλογα και με τις ε, συνθήκες γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι ό,τι έχετε από τη Ρωσία είναι fake news και όλα τα άλλα είναι καλές ειδήσει. Εμένα με απασχολεί. Ε, με απασχολεί αυτό το φιλτράρισμα, το μπλοκάρισμα. Αυτό είναι λογικό και πραγματικά Όσον αφορά τις ψευδείς ειδήσει, ε, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους ε, συμπολίτες μας, να τους δώσουμε πολύ καλά εργαλεία για το τι είναι ψευδή είδηση και τι όχι και αν τους εκπαιδεύσουμε τότε δεν θα είναι απαραίτητο να φιλτράρονται οι ειδήσει. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι φυσικός και πληροφορικάριος. Έχω μερικές ερωτήσεις για σας κύριε Κριστιανίνη. Είπατε ότι η πρόβλεψη μιας ε, συμπεριφοράς, ανθρώπινης ε, συμπεριφοράς, ε, βασίζεται σε προηγούμενη συμπεριφορά και ότι αυτό γίνεται. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το ποσοστό, η πρόβλεψη αυτή μιας επερχόμενης συμπεριφοράς ενός ανθρώπου να είναι σωστή. Γιατί αν αυτό το ποσοστό είναι 20%, δηλαδή 20% σωστή πρόβλεψη, τότε είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Τώρα, μια δεύτερη ερώτηση για το Google και το Facebook. Εγώ τα χρησιμοποιώ, έτσι, και είμαι πολύ ικανοποιημένη που τα χρησιμοποιώ. Αλλά ποτέ δεν λαμβάνω υπόψη πληροφορίες στις αποφάσεις που παίρνω εγώ. Δηλαδή, τις πληροφορίες που διαβάζω στο Google και στο Facebook δεν τις χρησιμοποιώ για τις αποφάσεις μου, γιατί δεν ξέρω τι αξιοπιστία έχουν. Για το Google είπατε ότι γνωρίζουμε ας πούμε κάποιες ιστοσελίδες, κάποια site που είναι αναξιόπιστες. Πώς μπορούμε, πώς μπορώ εγώ ας πούμε που κάνω μια έρευνα στο ίντερνετ να αποκλείσω ιστοσελίδες που είναι αναξιόπιστες. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εσείς ίσως το ξέρετε. Τώρα για το Facebook. Όλοι οι τρομοκράτες είχαν προφίλ και λογαριασμούς στο Facebook. Και μου είπανε, όταν είπα διαγράψτε τα ας πούμε, μου είπαν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε, δεν ξέρουμε ότι είναι τρομοκράτες. Όχι, το ξέρετε θα μπορούσατε να κάνετε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα στη βάση δεδομένων σας και θα μπορούσατε στο προφίλ Facebook να βάλετε ως υποχρέωση το σεβασμό των, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το... τη μη διάδοση του μίσους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι γίνεται. Uh, λοιπόν, όσον αφορά... Μισό λεπτό. Ε, την πρώτη ερώτηση θα απαντήσω που έχει σχέση με το αν ή μη ή αναξιόπιστε οι πληροφορίε που έχει σχέση και με αυτό που λέει προηγουμένω σχετικά με τον έλεγχο των γεγονότων. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με το πώ ε, θα ε, ετικετάρονται, πώ θα τοποθετούν ετικέτε σε συγκεκριμένα περιεχόμενα. Ε, τα μέσα κοινωνική δικτύωση, ξέρετε τι γίνεται, εκεί μοιάζουν όλα ίδια και δεν υπάρχει τρόπο να διαχωρίσει κανεί το αξιόπιστο από το αναξιόπιστο. Σωστή αυτή η κριτική ότι η ε, τεχνολογία είναι εξισωτική, ότι πράγματι θα πρέπει να βρούμε εργαλεία για να προσφέρουμε περισσότερες πληροφορίες και όταν ε, υπάρχει μια νέα πηγή ε, θα πρέπει κανείς να ξέρει αυτή πότε εμφανίστηκε, ε, χτες, μήπως ή υπάρχει εδώ και 100 χρόνια. Πράγματι αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες. Δεν είναι κακό να υπάρχει μια πηγή μόνο μια μέρα. Χρειαζόμαστε τέτοιου είδου εξέλιξη. Απλά είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τώρα για την τρομοκρατία θέλησα να ξεκαθαρίσω ότι κατά το παρελθόν οι εταιρείε του διαδικτύου ήταν πολύ επιφυλακτικέ στο να χρησιμοποιούν τη δική μα την τεχνολογία για να εντοπίζουν εκείνου που είναι επικίνδυνοι από το πρίσμα τη τρομοκρατία. Σκληρό βέβαια, δύσκολο και εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που κάνουν κακά πράγματα θα χρησιμοποιηθούν και αυτοί ε, τις υπηρεσίες της αγοράς, όπως το κάνουμε και εμείς, όλοι οι άλλοι. Αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, ε, παραδείγματο χάρη, ε, σε σχέση με την προπαγάνδα που γίνεται, να την αφαιρούμε και όταν υπάρχει μία αξιόπιστη απειλή, πράγματι να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές. Μπορούμε βέβαια να δούμε τώρα τι είναι αξιόπιστη απειλή και τι όχι. Πάντως, η άποψη της εταιρεία μας είναι ότι οφείλουμε να χρησιμοποιούμε την ευφυή τεχνολογία για να προστατεύουμε τους ανθρώπους, το δικαίωμά τους στη ζωή. Ε, στις 6 Δεκεμβρίου ο κύριος ε, Αβραμόπουλος οργανώνει εδώ μία συνάντηση ε, και εκεί θα δείξουμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να προστατεύονται οι άνθρωποι από τους τρομοκράτες. Και εγώ θα απαντήσω και τις δύο ερωτήσεις, αλλά επιτρέψτε μου να επανέλθω στην ερώτηση του κύριου Βερουλευτή για την ιδιωτική σφαίρα και τα κινητά. Ε, μπορείτε να αποφασίσετε μόνο σας μέσα στο κινητό ε, ποιες ειδήσει ε, θα είναι προσβάσιμες σε όλους και ποιες όχι. Υπάρχει το σχετικό app, υπάρχει ο έλεγχος και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για να προστατεύετε την ιδιωτική σας σφαίρα επίση, ε, σε άλλε ερωτήσεις και οι δύο κατ' ουσίαν ερωτήσατε την ίδια ερώτηση με άλλο τρόπο. Δηλαδή πώς ε, αποφασίζουμε το περιεχόμενο που προβάλλουμε και κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος ε, η λογοκροσία να είναι τελικά πρόβλημα. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας πω ότι υπάρχει η πρόθεση να βρούμε χρήσιμες πληροφορίες και να αναλαμβάνουμε όμως και τις ευθύνες μας. Ε, θέλω όμως να πω ότι τα αποτελέσματα τα λογοκρίνουμε γιατί κάνουμε ε, επιλογές ε, μέσα από μηχανές μάθησης, με αλγορίθμους. Αυτό δεν είναι λογοκρισία, δεν είναι ότι απομακρύνουμε το περιεχόμενο, Απλά λέμε ότι με βάση την έρευνα που κάναμε, ε, τα αποτελέσματα που σας δείχνουμε είναι και τα πιο χρήσιμα. Ανέφερα παραδείγματος χάρη ε, το, την περίπτωση του ολοκαυτώματος, όπου θελήσαμε να δείξουμε κατά πόσον αυτή η πηγή για την άρνηση του ολοκαυτώματος ήταν αξιόπιστη ή όχι. Και το κάναμε αυτό εξετάζοντας συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Η απάντηση είναι ότι όχι, δεν υπάρχουν αξιόπιστα site επ' αυτού του θέματος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αν ψάχνει κανείς ε, να βρει κάτι σχετικά με την άρνηση του ολοκαυτώματος, ε, δεν μπορεί να βρει κάτι. Ε, εμείς αφαιρούμε από τους ε, έρευνες περιεχόμενο μόνο εφόσον υπάρχει δικαστική απόφαση. Μετά από δικαστική απόφαση. Εμείς δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε και δεν το κάνουμε, απλά χρησιμοποιούμε κάποια μηνύματα και αλγορίθμους που νομίζω ότι απαντούν την ερώτησή σας για το πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ότι το περιεχόμενο που έχουμε δείξει είναι χρήσιμο για κάποιον και, άλλο, και όχι για άλλον. Αυτά είναι τα μηνύματα που έχουμε να χρησιμοποιήσουμε, αυτά είναι τα σημειάλα και ε, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να δώσουμε και τις ε, πιο χρήσιμες ε, πληροφορίες. Ευχαριστούμε, Τζον. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ε, δεν έχουμε πια άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε που μείνατε και συμμετείχατε σε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ευχαριστώ επίσης και όλα τα μέλη του πάνελ. Και πριν δώσω το λόγο ε, στην κυρία Καλή, στην πρόεδρο της Επιτροπής ΣΤΟΑ, ε, θέλω να πω ότι μάθαμε πάρα πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί. Ελπίζω όμως ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι θα βρούμε λύσεις σε σημαντικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας και θα συνεχίσουν να την απασχολούν τις επόμενες δεκαετίες. Σας ευχαριστώ πολύ. First of all, I want to invite uh, Vice Chair of STOA, Mr. Paul Rubik. Κύριος Πολ Ρούμπικ, αντιπρόεδρος της ΣΤΟΑ uh, και ο αντιπρόεδρος Ραμόν Λουίς Βαρκαρέλ, υπεύθυνος της ΣΤΟΑ, θα έρθουν εδώ στο βήμα. Σας ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε. Ήταν θαυμάσια η συζήτηση. Ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής είναι η επικοινωνία. David, έχεις ένα πολύ δύσκολο καθήκον, είχες ένα πολύ δύσκολο καθήκον σήμερα. Εσύ και σε ευχαριστώ για αυτό. Ε, και ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές. Πολ ε, ε, just... και ο Αντιπρόεδρος θα έρθουν στο βήμα. Ακόμα 10 λεπτά. Και μετά υπάρχει ένα κοκτέιλ. Εκεί μπορείτε να ρωτήσετε όλα και να σας απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που δεν σας απαντήθηκα στο ισόγειο. Θα ακολουθήσετε τους βοηθούς μας και θα σας οδηγήσουν στο συγκεκριμένο χώρο. Υπάρχει ένα hub ε, με μηχανισμό παρατηρητηρίου ε, για θέματα επικοινωνία, ε, επικοινωνίας και επιστήμης. Ο κύριος Ζούμπι θα πει δύο λόγια και μετά ο Αντιπρόεδρος θα κλείσει την ε, θαυμάσια αυτή ετήσια εκδήλωση της ΤΟΑ. Σε μια συνάντηση για την ε, ασφάλεια υπήρχε ένας ειδικό ε, που φτιάχνει λογισμικό για την κυβερνοασφάλεια. Αν θες να ξέρεις, είπε, πώς θα γίνεις ασφα... ασφαλής από τις νέες τεχνολογίες και την ε, τεχνητή νοημοσύνη, ε, η απάντηση που... και θες να είσαι 100% ασφαλής, μία είναι η απάντηση. Να μην τη χρησιμοποιεί. Εμείς θέλουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, αλλά να τη χρησιμοποιούμε με προσοχή και θέλουμε ως πολιτικοί να προστατεύεται η ιδιωτική σφαίρα των πολιτών μας. Γι' αυτό ακριβώς ήταν πάρα πολύ η σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ την Εύα Καϊλή και χαίρομαι που κάθομαι δίπλα σε έναν μηχανικό. Ε, γιατί στην πολιτική... Ε, δεν συμβαίνει κάθε μέρα αυτό. Σήμερα διαμορφώνουμε πράγματα που θα πάρουν μορφή μετά από 30 χρόνια. Του χρόνου θα έχουμε την Προεδρία για μια ομάδα που κάνει αξιολόγηση μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια για θέματα τεχνολογίας ε, θέλουμε να βγούμε και σε πιο διεθνές επίπεδο. Η συνεργασία επιστημών και πολιτικών είναι πολύ σημαντική και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην τεχνολογία. Στη ΣΤΟΑ ξέρουμε ότι η κινητικότητα, ας θα είναι ένα από τα μεγάλα θέματα του μέλλοντος. Όχι μόνο με τα bits και τα byte, αλλά κινητικότητα περιεχομένου, ε, ανθρώπων, αγαθών, κιλοβατόρων, Και προφανώς εκεί θα ανακύψει και το θέμα των πόρων. Τι είναι ε, μια τυποποίηση 5G, 6G. Ε, πώς έχουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Και πώς θα έχουμε και την ενόραση για να προβλέψουμε τι επίπτωση θα έχουν οι διάφορες τεχνολογίες. Θέλουμε να βγούμε από τη στρατηγική της, του κατακαιρματισμού. Ο καθένας από, από είναι ένα τέτοιο ας πούμε, κομμάτι γνώσης, μια ψηφίδα γνώσης. Το θέμα είναι πώς αυτές οι ψηφίδες θα φτιάξουν ένα όλο. Ε, το θέμα δεν είναι μόνο ποιότητα, δεν είναι μόνο ποσότητας, δεν είναι μόνο χρόνου. Έχουμε πολλές δραστηριότητες όπου η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλγόριθμοι θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. όχι μόνο για να είμαστε σίγουροι ποιος θέλει ποια πληροφορία, αλλά να σας δώσουμε με υπευθυνότητα τις πληροφορίες που θέλετε, που σας ενδιαφέρουν. σε εσά θα δώσουμε τι χι πληροφορίε, ενώ σε κάποιον άλλο που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για αυτέ τι πληροφορίε, δεν έχει κανένα νόημα να του δίνουμε τι ίδιε ακριβώ πληροφορίε, αφού δεν τον ενδιαφέρουν. Κάνω μια μεγάλη συζήτηση εδώ στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες. Τρεις εβδομάδες το μήνα είμαστε στις Βρυξέλλες, μία εβδομάδα το μήνα είμαστε στο Στραβούργο. Έχουμε πολλές υποδομές πολύ... και πολλοί κόσμος ας πούμε, μας ρωτάει γιατί ξοδεύεται τόσα χρήματα ας πούμε, και αφήνεται άδειο το κτίριο του Στρασβούργου. Ε, Οι Γάλλοι είδαμε ότι είναι πολύ καλή στην τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Ε, έχουμε πολύ καλή συνεργασία εμείς Γερμανοί με την, ε, μέσω της ΑΡΤΕ. Ε, πολύ καλή επίσης συνοριακή συνεργασία με τη Γαλλία. Δημιουργούμε ένα κέντρο που μπορεί να ε, δώσει νέας μορφής πληροφορίες. Ε, κάποτε Ή, λέγαμε ότι η πολιτική είναι καλύτερη, δημοσιογράφη, ειναι καλύτερη από τους δημοσιογράφους. Ε, ίσως τώρα αλλάζουν αυτά τα πράγματα χάρη στις ε, νέες πλατφόρμες. Οι δημοσιογράφοι θα γίνουν καλύτεροι από τους πολιτικούς. Είμαι σίγουρος ότι είμαστε στην απαρχή της πλατφόρμας αυτής. Θα υπάρξουν πάρα πολλές εξελίξεις. Θέλουμε να είμαστε στους προμαχώνες. Πώς ε, αντιμετωπίζουμε την ε, λογική της, ε, του κατακαιρματισμού και σπάμε τον κατακαιρματισμό. Έχουμε τις υποδομές στο στις Βρυξέλλες, αλλά και στο Στρασβούργο έχουμε εξοπλισμό. Μαζί με την ΕΒΑ ξεκινήσαμε ε, στα πλαίσια της Επιτροπής Προπολογισμών να βρούμε, ψάξαμε να βρούμε την νομική βάση για να ασχοληθούμε με θέματα ε, έψιλων. Βρήκαμε κάποια λεφτά, μπορούμε να τα κάνουμε μελέτες ε, για να παράγουμε τη σωστή γνώση και να εκπαιδεύσουμε όχι μόνο τους βουλευτές και το προσωπικό μας του Κοινοβουλίου, ε, όχι μόνο τους οργανισμούς των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, αλλά θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, μια πολύ καλή, ένα καλό team που θα συνεργάζεται με το Κοινό Κέντρο Ερευνών ε, τη στιγμή που ξοδεύουμε δισεκατομμύρια ευρώ ε, σε ερευνητικά προγράμματα. Ε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή τη γνώση που παίρνουμε ε, και μπορούμε να την ε, καθοδηγήσουμε από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο και τις μεγάλες εταιρείες. Ε, πώς θα επικοινωνήσουμε με νέους τρόπους, ε, πώς θα χρησιμοποιήσουμε ας πούμε τα infographics για να ανοίξουμε τις κοινωνίες μας. Ξεκινάμε αυτή τη διαδικασία από 1η πρώτη 18. Θα έχουμε ε, αυτό το συμβουλευτικό όργανο στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με διανοητές, με εμπειρογνώμονες, ούτως ώστε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις πληροφορίες και πώς μπορούμε στα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους να τους δώσουμε τα στοιχεία για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα παγκόσμιο κέντρο που καλεί κόσμο από όλες τις χώρες, ούτω ώστε να πούν την άποψή τους, να αποφεληθούμε από τις γνώσεις τους και ακριβώς αυτό που κάναμε σήμερα χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αυτή την ανοιχτή συζήτηση, να λέμε ότι αυτό είναι θετικό, αυτό είναι αρνητικό, αυτό είναι πιθανό, αυτό είναι απίθανο να γίνει. Φυσικά δεν θα έχουμε πάντα τις ίδιες απόψεις σε όλα τα θέματα, αλλά με αυτόν τον τρόπο η πολιτική είναι πλούσια. Αλλά σας λέω ότι η ΣΤΟΑ δεν, είναι, δεν υπάρχει για να παίρνει αποφάσεις. Εγώ συχαίνομαι τις αποφάσεις. Μ' αρέσει να έχω εναλλακτικέ λύσεις, να τις δημιουργώ. Να βλέπω πώς αλλάζουν και να βλέπω ποιε είναι οι επιπτώσει των διαφόρων εναλλακτικών. Μερικές φορές υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού, μερικές φορές δεν υπάρχει. Αλλά με χαρά σας αναγγέλλω εδώ και τώρα ότι θα υπάρξουν αυτέ οι συναντήσεις. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μα και βοηθήστε μα να καλλιεργήσουμε αυτή την ιδέα, να την περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Τώρα απλώς ξεκινήσαμε. Αυτή η συνεργασία επιστήμης ΜΜΕ είναι σημαντικό να γίνει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τελεσφορήσει αυτή η ιδέα. Και ο κύριος Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε της ΤΟΑ. Ευχαριστώ Εύα Καϊλή Και ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Πολ Ρούμπικ. Κυρίες και κύριοι. Και για μένα πρέπει να σας πω ότι είναι απίστευτη η ικανοποίηση που φτάσαμε σε αυτή τη φάση αυτής της ετήσιας διάσκεψης. Ακόμα μία φορά ήταν επιτυχής και σε ό,τι αφορά την προσέλευση όπως βλέπετε, αλλά και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο. Είναι υποχρεωτικό καταρχάς να ευχαριστήσω όλη την ομάδα της ε, Επιτροπής μας για τις ε, επιστημονικές και τεχνολογικές ε, επιλογές που έκανε μια θαυμάσια δουλειά ούτω ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτή η διάσκεψη. Ως Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, υπεύθυνο για την ΣΤΟΑ στο Προεδρείο, θα συμμετάσχω, όχι πάντα, αλλά όσο μπορώ πιο συχνά στις συζητήσεις για τα θέματα εφαρμογών των νέων τεχνολογιών. Το σίγουρο είναι ότι το περιεχόμενο των συζητήσεων στις οποίες ε, παρευρεθήκατε σήμερα πραγματικά ήταν με ενέπνευσε θα έλεγα. Οι συζητήσεις, οι παρουσιάσεις μας καλούν να πάμε πιο πέρα από το όριο της σκέψης μας και μας καλούν επίσης ε, στη σύνεση και στην προσοχή είναι το καλύτερο δώρο για ένα που μπορεί να κάνει ένας ομιλητέ. δηλαδή να ξυπνήσει το ενδιαφέρον του κοινού του. Και είμαι σίγουρος ότι οι προλαλήσαντες ακριβώς ε, αυτό έκαναν, ξύπνησαν το ενδιαφέρον σας. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη διάσκεψη, εδώ στην αίθουσα, αλλά και όσοι την παρακολούθησαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στην ε, παρέμβαση του κυρίου Χριστιανίνη, ο οποίος εξήγησε πώς η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλγόριθμοι διαχειρίζονται ροές πληροφοριών χωρίς να το καταλάβουμε εμείς. Δεν εκπλήσω κανέναν όταν λέω ότι στις 21 Νοεμβρίου του 2017, σήμερα δηλαδή, προσπαθούμε να προωθήσουμε πολιτικές ε, στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τους αλγόριθμους πληροφοριών. Ακούσαμε δυστυχώς πάρα πολλές κακές και ανησυχητικές ειδήσεις τα τελευταία χρόνια. Είδαμε ας πούμε πως ξένες δυνάμεις, χάρη στο, στην κυριαρχία που έχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσω ανορθόδοξων τεχνικών κατάφεραν να επηρεάσουν ας πούμε, δημοκρατικές διαδικασίες μεγάλων χωρών. Και να επηρεάσουν ε, επιταχύρω τα αποτελέσματα εκλογικά. Το ίντερνετ έχει αντικαταστήσει πολλά πράγματα του παρελθόντος. Ε, έχει αντικαταστήσει τα, τα χαρακόμματα του παρελθόντος. Ε, και τα πυρομαχικά ποια είναι του ίντερνετ, η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς ειδήσει, η επιτούτου παραπληροφόρηση. Μια παραπληροφορημένη κοινωνία είναι μια κοινωνία έτοιμη για να την εκμεταλλευτείς. Οι αλγόριθμοι όμως από την άλλη δίνουν και τεράστιες ευκαιρίες για τα συστήματα δημιουργίας, διαχείρισης, διάδοσης πληροφοριών ε, για θέματα υγείας, για την αναζήτηση εργασίας, όπως είπαν κάποιοι ομιλητέ. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να μελετούμε πώς θα εξασφαλίσουμε ότι εμείς είμαστε εκείνοι που ελέγχουμε τους αλγοριθμούς μας και όχι το αντίθετο. Και ας στάσουμε στο θέμα της ε, αδιαφάνειας των ε, μέσων κοινωνικών, ε, κοινωνικής δικτύωσης μέσω των αλγορίθμων τους. Ακούσαμε διάφορες περιπτώσεις διακρίσεων, ας πούμε, που οδηγούν και στο μίσος ή που αναμοχλεύουν το μίσος με τη διάδοση ε, ψευδών ειδήσεων. Η ευθύνη δεν είναι μόνο στους α, αλγόριθμους μερικές φορές ε, επίτηδες αφήνουμε αυτές τις ειδήσει και, και το θέμα πάει πέρα από τον έλεγχο που έχουμε στους αλγορίθμους. Είναι και θέμα δηλαδή πρόθεσης. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν μοντέλα διαφάνειας, ούτω ώστε να έχουμε μηχανισμούς επαλήθευσης των λογαριασμών. και επίσης να ελέγχουμε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις με τη χρήση αλγορίθμων. Πέρα από διάφορους υπολογισμούς που κάνουμε, θα πρέπει να δούμε και κάποια άλλα θέματα ε, διοντολογικής φύσεως. Ακόμα πιο περίπλοκο είναι θα πρέπει ε, η απόφαση που θα πάρουμε για το επίπεδο διαφάνειας που θέλουμε να έχουμε. Επίσης, τι θέση πρέπει να έχει όλα αυτά ο χρήστης και πώς εκείνος ας πούμε, μπορεί να προτάξει τις ε, προτιμήσεις του σε ένα σύστημα το οποίο αποφασίζει για το ποιες είναι οι δικές του προτιμήσεις. Για λογαριασμό του αποφασίζει. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι το να υπάρχει ένα επιστημονικό κέντρο για να εκπαιδεύει τους πολίτες. Κυρίες και κύριοι, πρωτοβουλίες όπως η σημερινή αποτελούν χωρίς καμία αμφιβολία ένα βήμα προς το να κάνουμε την επιστήμη όσο και όλο και πιο προσιτή στους πολίτες, πιο εκλαϊκευμένη, αλλά και πραγματική. Θα πρέπει να έχουμε σχέση ανάμεσα στις κοινωνικές διεργασίες και τα κοινωνικά δρόμανα και στις επιστημονικές εξελίξεις. Αυτό είναι ο βασικός και φιλόδοξος στόχος της ΣΤΟΑ. Θέλω να τελειώσω ευχαριστώντας την πρόεδρο της Επιτροπής και τον αντιπρόεδρο, καθώς και τους υπόλοιπους συναδέλφους να παρτίζουν, για τη δέσμευση, την ε, ανάμιξή τους, ε, προκειμένου να τελεσφορήσει αυτή η εκδήλωση. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω την ε, προσπάθεια που κάνουν οι υπηρεσίε επικοινωνία και διερμηνία. Χωρί αυτού δεν θα ήταν δυνατή η σημερινή εκδήλωση. Σα ευχαριστώ ακόμα πάρα πολύ και εμεί σα ευχαριστούμε. Και σας προσκαλώ στο κοκτέιλ το οποίο θα λάβει χώρα στο σαλόνι των Ευρωβουλευτών στο κτίριο Αλτιέρο Σπινέλη. Ακόμα μια φορά σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για τη συμμετοχή σας. Γεια σας. While you're packing, I will just thank Zolt, Michalis, Philippe, Gerasimos, Live,